Um, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω καμία, κανέναν να διαφωνεί. Οπότε θεωρώ ότι εγκρίνεται. Δυστυχώς έχω κάποιες ανακοινώσεις πρώτα. Όπως ξέρετε, 27 Οκτωβρίου ο πρόεδρος Μπαρός ανακοίνωσε αλλαγές στα χαρτοφυλάκια των Επιτρόπων Ρεν και Σεμέτα και οι δύο αυτές αλλαγές είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας και σύμφωνα με το άρθρο 106,6 του κανονισμού και τα παραρτήματα πρέπει να γίνει άλλη μια ακρόαση χωρίς ψηφοφορία για τους επιτρόπους αυτούς. Μπορώ να σας πω πως έχουν προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου το απόγευμα οι ακροάσεις και θα σας δώσουμε λεπτομέρειες. Το γεγονός πως ο κύριος Ρεν βρίσκεται εδώ πέρα σήμερα είναι συμπτωματικό, δεν έχει σχέση με τις νέε του αρμοδιότητε. Για την οδηγία MIFID θα γίνει μια δημόσια ακρόαση την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30. Μια ημερομηνία που δεν είναι στο πρόγραμμά μας, οπότε είναι μια επιπρόσθετη ημερομηνία, 5 Δεκεμβρίου 3 η ώρα, για την εγγύηση καταθέσεων για τον τριμερή διάλογο Είχαμε δεύτερο τριμερή διάλογο στις 26 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια του Στρασβούργου και οι διαπραγματεύσεις έφτασαν σε αδιέξοδο καθώς η Πολωνική Προεδρία μας είπε πως είναι άκαμπτο το Συμβούλιο για το επίπεδο στόχου των ε, κονδυλίων και υπήρχε περιορισμένη ευελιξία για την περίοδο πληρωμής Οπότε σκοπεύουμε να γίνει η επόμενη συνάντηση πριν από την επόμενη συνεδρίασή μας 15 Νοεμβρίου και αν εξακολουθούμε να μην συμφωνούμε θα σκεφτούμε την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Όσον αφορά το ζήτημα ΣΥΠΕΡ, είχαμε το δεύτερο τριμερή διάλογο στις 26 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Όλα τα βασικά σημεία έχουν καλυφθεί, έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος ένα ενημερωμένο έγγραφο με συμβαστικής λύσης έχει δοθεί σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις κλειδιά που πρέπει να ε, ληφθούν ακόμα, μεταξύ των οποίων και η ημερομηνία λήξης για τα συστήματα νη ΣΥΠΕΡ. Ελπίζουμε όμως ακόμα σε συμφωνία τον Νοέμβριο η επόμενη συνάντηση προγραμματίζεται για τις 16 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις. Οπότε χαίρομαι τώρα που θα περάσουμε στην δημόσια κρόση. Όπως είμαι σίγουροι πως θα ξέρετε αυτή τη στιγμή η καιρή είναι δύσκολη. Έχουμε τον κύριο Ροστόφσκι, πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ και τον Όλη Ρέναντι, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών. μας ενημέρωσε το γραφείο των Χέρμαν Φανρόμποη και Τζούλιο Τρεμόντι πως είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις και δεν μπορούσαν να έρθουν. Και βεβαίως αναμένουμε την πλήρη εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την οικονομική διακυβέρνηση και βεβαίως και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής, οπότε θα απευθύνω μία επιστολή στον κύριο Φανερόμπα για να κάνουμε ένα διάλογο μαζί του. Επίσης θα είδατε πως βρίσκεται εδώ πέρα και ο κύριος Γιώργη Ματόλσκι, πρώην πρόεδρος ε, του ε, Συμβουλίου Εκοφήν, ε, ο οποίος θα έπρεπε να είναι εδώ, αλλά και αυτός είχε μία ξαφνική υποχρέωση. Και βεβαίως λόγω και του Eurogroup το οποίο συνεδριάζει οι ομιλητές θα χρειαστεί να φύγουν λίγο νωρίτερα. Οπότε θα τα δούμε τα πράγματα αναλόγως με το πώς θα κυλήσουν. Στον κύριο Γιάνν Βίνσεν να πληρώνει ο υφυπουργός του. Λοιπόν, ο κάθε ομιλητής θα έχει πέντε λεπτά για να κάνει τις παρατηρήσεις του. Θα σας ακούσουμε και τους δύο και μετά νομίζω θα ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις για να μπορέσετε να απαντήσετε πριν ε, φύγετε βεβαίως. Όταν είχαμε κανονίσει την ακρόαση δεν ξέραμε βεβαίως πως θα συνέπιπτε ε, με... με τη συγκυρία αυτή. Οπότε θα δείξουμε κάποια κατανόηση. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη γιατί σε λίγο θα πρέπει να φύγω. Αλλά ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε όσο δυνατό περισσότερες ερωτήσεις και να απαντήσω όσο το δυνατό περισσότερες μπορώ. Μια και είναι η πρώτη φορά που έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την έκριση του πακέτου των έξι νομοθετικών ε, μεταρρυθμιστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω και είμαι σχεδόν πεπισμένος ότι θα αποφύγουμε επανάληψη των ε, ίδιων προβλημάτων. Και χαίρομαι ειλικρινά που καταφέραμε να καταλήξουμε συμβαστική λύση προκειμένου να γίνει δεκτό αυτό το εξάπτυχο πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Νομίζω ότι καλό είναι να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να εκφράσουμε την ευαρέσκειά μας ε, για τη σημασία αυτής της συμφωνίας. Έγιναν πολλά σημαντικά πράγματα, ήταν πολλά τα επιτεύγματα και χάρη στη συνεργασία και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταφέραμε και καταλήξαμε σε αίσιο πέρας, ε, σε μια συμβαστική λύση. Θα ήθελα να πω Χαίρομαι για την ευκαιρία που δίνεται στην ε, Πολωνική Προεδρία να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τις εμπειρίες που συγκεντρώσαμε από την εφαρμογή αυτού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ήταν πολύ εντατική αυτή η έναρξη αυτού του εξαμήνου και η αξιολόγηση της ε, διαδικασίας δεν έχει ούτε καν ξεκινήσει, όχι ολοκληρωθεί. Εν πάση περιπτώσει, παρόλο που βρισκόμαστε σε πολύ εισαγωγικό στάδιο, είναι χρήσιμο που έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων γι' αυτό. Εν είδη εισαγωγή, θα ήθελα να προβώ σε μια σύντομη ανάλυση της κατάστασης, γιατί η τρέχουσα κατάσταση θα επηρεάσει και τις μελλοντικέ αποφάσεις, τις αποφάσεις που θα χρειαστεί να λάβουμε και για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Όπως ξέρετε, η κρίση δημόσιου χρέους ε, ε, ε ενέχει τον κίνδυνο της ε, ε και τραπεζικών κρίσεων και μπορούμε να βρεθούμε σε ένα αρνητικό σπιράλ που οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ θα αφιβάλλουν όλο και περισσότερο για τη δυνατότητα των χωρών μελών να εξυπηρετήσουν το χρέο του. Και αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες στις τράπεζες που έχουν στον ισολογισμό τους ε, ε, μετοχές, ε, ομόλογα μάλλον δημόσιο χρέου. Οπότε θα υπάρξουν προβλήματα στη χρηματοδότηση των τραπεζών και στη διατραπεζική αγορά. Έχουμε διαπιστώσει τέτοιου είδους προβλήματα και μάλιστα αυτό το επισήμανε και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στο παρελθόν ε, οι τραπεζικές κρίσεις ε, είχαν οδηγήσει σε σοβαρές κρίσεις και στην πραγματική οικονομία. Και η κρίση που ξεκίνησε το 2008 ήταν μια χρηματοπιστωτική κρίση που στη συνέχεια μετατράπηκε σε κρίση και της πραγματικής οικονομίας. Η παρούσα κρίση ξεκίνησε στις αρχές του 2010, ήταν αρχικά κρίση δημοσίου χρέους και μετατράπηκε στην πορεία σε κάποιο βαθμό, όχι πλήρως ακόμη και χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά έχει τη, τη πιθανότητα να μετατραπεί σε κρίση και το χρηματοπιστωτικό τομέα. Δεν έχει ακόμη μετατραπεί σε τέτοια χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά περιέχει τέτοιο, τέτοιες δυνατότητες, τέτοιο δυναμικό. Και παρόλο που δεν είναι κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ήδη με ρυθμούς γίνεται κρίση της πραγματικής οικονομίας και όλοι συμφωνούμε ότι η κατάσταση είναι δεινή, σοβαρή και θα έχει βαθύτερες και κατά πάσα πιθανότητα μακροπρόθεσμες συνέπειες στην απασχόληση, την ανάπτυξη και την φτώχεια. Και νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς είναι η καταλληλότερη στιγμή σήμερα να εξετάσουμε τα διάφορα μέτρα που προσπαθήσαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβουμε για να αντισταθμίσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτές τις δυσκολίες, να δημιουργήσουμε ένα αντίβαρο. Και ένα τμήμα αυτών των προσπαθειών ε, ήταν και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χολιράν. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να ανταλλάξαμε απόψεις ε, σχετικά ε, με αυτό το, ε, την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πριν την θέση σε ισχύ της δέσμης των έξι μέτρων. Ευχαριστώ πολύ και για τις γραπτές ερωτήσεις που μου έχετε υποβάλει. Είναι πραγματικά σημαντικό που βλέπω ότι το Κοινοβούλιο εστιάζει πάνω σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι πολύ σωστά όλα αυτά που είπε ο κύριος Ροστόφσκι όσον αφορά την ολοκλήρωση ε, του πακέτου μετά από πάρα πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Θα ήθελα μάλιστα να σας συγχαρώ όλους ε, και ε, προσδοκούμε ε, ειλικρινά γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου τη θέση ισχύ της δέσμης αυτής. Θεωρώ ότι αυτή η δέσμη ε, μπορεί να ενδυναμώσει την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως δε στην Ευρωζώνη και αυτό ε, για το καλό της οικονομικής σταθερότητας, της αηφόρου ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορώ να πω ότι θα πρέπει να είστε ήσυχοι ότι δηλαδή θα χρησιμοποιηθούν από την πρώτη κιόλας μέρα όλα τα εργαλεία ε, αυτής της δέσμης μέτρων. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο βεβαίως άμεσα συνδέεται με την δέσμη ε, των ε, έξι μέτρων και θα εξηγήσω την άποψή μου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την εμπειρία αυτή σε λίγο. Αλλά θα ήθελα να πω δύο λόγια σχετικά με την σημερινή συνάντηση του Eurogroup πριν ασχοληθώ με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Έχουμε, είχαμε πολλά ε, σημαντικά ζητήματα, την Ελλάδα, την Ιταλία, την ε, ε, ενίσχυση ε, του FSF και των εργαλείων του πολλά ζητήματα ε, τα οποία βεβαίως ε, συνδέονται και με τις ε, συζητήσεις που έγιναν στις Κάνες στα πλαίσια του G20 και τη συνεργασία και τις συνομιλίες με το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο. Η σημερινή συνεδρίαση λοιπόν λαμβάνει η χώρα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη συγκυρία μετά από τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις οι οποίες άλλωστε δεν έχουν ολοκληρωθεί στην Ελλάδα. Ε, στα πλαίσια της G20 στις ε, Κάνες την προηγούμενη εβδομάδα πολύς χρόνος εξοδεύτηκε και πολλή συζήτηση έγινε για την Ευρωζώνη. Πολλές συμβουλές ακούσαμε και στήριξη ε, πολύ από τους εταίρους μας η G20 καλωσόρισε τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη διάσκεψη κορυφή, στη Σύνοδο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Ελλάδα να ενδυναμώσει και το τραπεζικό της ε, σύστημα και ε, να αποφευχθεί εν πάση περιπτώσει η μόλυνση και η μετάδοση ε, στις άλλες χώρες και οπωσδήποτε να γίνει πιο δυνατή η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη. Αποφάσισε ο Έλληνας Πρωθυπουργό Γιώργος Παπανδρέου την προηγούμενη εβδομάδα ε, να διεξάγει δημοψήφισμα ε, σχετικά με ερώτημα, δηλαδή σχετικό ε, με το κατά πόσον συμφωνούν οι Έλληνες με την συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου, η οποία είχε όμως γίνει αποδεκτή ήδη την 26η Οκτωβρίου στην Σύνοδο Κορυφής την προηγούμενη εβδομάδα και τις προηγούμενες μέρες ε, είδαμε πολλές εξελίξεις στην Ελλάδα. Πάντως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εμείς παραμένουμε δεσμευμένοι στην υπόθεση της Ελλάδας καθώς επίσης και σε αποφάσεις 26 Οκτωβρίου αλλά θα πρέπει και η Ελλάδα να ε, μην αποκλίνει από αυτές τις αποφάσεις επί των οποίων έχει δεσμευτεί. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο έτσι ώστε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Ε, γίνονται διεργασίες ε, για κυβέρνηση εθνικής ενότητας και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει ε, μια ανάνεψη της εμπιστοσύνης καθώς επίσης και ανάληψη των ευθυνών της 20 που απορρέουν από τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου και ξέρω ότι ο Υπουργός Οικονομικών έρχεται στις ε, Βρυξέλλες και οπωσδήποτε θα μας πει νέα στο Eurogroup, στη συνεδρίαση που θα έχουμε σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Σχετικά με την Ιταλία, Πολλά, πολλής λόγος έγινε για την Ιταλία στα πλαίσια ε, της ε, συνάντησης των G20 ε, λόγω των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει και λόγω της τεράστιας αύξησης των spreads που είδε η Ιταλία την προηγούμενη εβδομάδα έχει αναλάβει δεσμεύσεις έτσι ώστε να εξηγιάνει τα οικονομικά της ε, και ε, βεβαίως ε, να έχει αναλάβει δεσμεύσεις σχετικά με, την, με το ευρωπαϊκό εξάμεινο και την ευθυγράμμιση της χώρας αυτής με τις αρχές του ευρωπαϊκού εξαμήνου λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα διορθωτικά προβλήματα της Ιταλίας για να δειχθεί μάλιστα έτσι περαιτέρω η αποφασιστικότητά της, ε, ε, της Ιταλίας εννοώ, ε, στον δρόμο αυτό έχουν αναλυφθεί νέες συζητήσεις και θα υπάρξει εποπτεία της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης στην Ιταλία έτσι ώστε να υπάρξει συγκεκριμένη και τελική αξιολόγηση. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, στην πράξη το ευρωπαϊκό εξάμεινο υλοποιείται πλέον μέσα σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Θα ήθελα να καλύψω ορισμένα κεντρικά ε, ζητήματα. Πρώτα υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την εθνική ε, αντιμετώπιση, εθνική αντίδραση μάλλον, ε, σε σχέση με την εθνική κυριαρχία και παρεμφερή ε, ζητήματα. Βεβαίως Καμία χώρα δεν μπορεί να είναι απολύτως σύμφωνη ή ευχαριστημένη όταν της δίνονται ε, συμβουλές. Το ζητούμενο πάντως είναι να υπάρξει μία εξάντε ε, δημοσιονομική εποπτεία έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι ε, πολύ καλύτερα. Είναι γεγονός ότι είναι σχετικός ο ενθουσιασμός, ο οποίος βεβαίως δεν έτυχε καθολικής έτσι, από τα εθνικά κοινοβούλια γιατί ακούγεται διαρκώς ότι οι Βρυξέλλες προσπαθούν ε, να ε, πάρουν ένα κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας ε, κλπ. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να καθησυχάσω όλο τον κόσμο και τα εθνικά κοινοβούλια. Είναι γεγονός ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να κατανοήσουν ποιοι είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες ε, και τα ίδια τα εθνικά κοινοβούλια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν εκ των προτέρων δεχτεί να σέβονται τους κανόνες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και ε, βεβαίως εδώ και μέσα από τον διακυβερνοβουλευτικό διάλογο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Λάμπερτς και στην ε, ομάδα των ε, Πρασίνων. Ε, πραγματικά ελπίζω ότι η μελέτη η οποία εκπονήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες θα διαβαστεί από όλους και σε όλες τις πρωτεύουσες. Είναι πολύ σημαντική εργασία. Επίσης, to η δημοκρατική ε, λογοδοσία είναι πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτό λοιπόν εμείς στηρίζουμε τον διάλογο. Οι συζητήσεις δεν θα λαμβάνουν πλέον χώρα και κλεισμένων των θυρών. Θα πρέπει να γνωρίζουν ε, όλοι τα τεκτενόμενα ε, και να γνωρίζουν όλοι τι διαμείβεται. Και ευελπιστώ λοιπόν ότι ο οικονομικός διάλογος θα έχει μόνο θετική επίπτωση. Δεν έχω πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μου, αλλά θα ήθελα να πω ακόμα κάτι. Να αναφερθώ δηλαδή στην δεύτερη ομάδα ερωτήσεων. Ε, στην ουσία να αναφερθώ στον ε, στρατηγικό αντίκτυπο της, ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση να κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση βασιζόμενη σε συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά την εθνική στρατηγική. Θα ήθελα ας πούμε να σας πω ότι η Ισπανία π.χ έχει ακολουθήσει τις εξειδικευμένες ε, ε, συστάσεις σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και πρέπει να πούμε ότι η χώρα αυτή τα πάει μάλλον καλά ε, παρά τις μεγάλες αλλαγές που έχει υποστεί η οικονομία της και το ποσοστό ανεργίας κτλ. Ε, η Σάρων έλεγε προηγουμένω ότι ενδεχομένως ε, θα μπορούσα να επανέλθω τον Ιανουάριο για περαιτέρω συζήτηση στην Επιτροπή σας, έτσι ώστε να συζητήσουμε περαιτέρω τον πολιτικό αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, για τον Ιανουάριο βεβαίως θα ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Θα ολοκληρώσω λοιπόν λέγοντας ότι ελπίζω ότι μέσω των παρατηρήσεών μου θα έχετε κατανοήσει όλοι ότι η δέσμευσή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θεωρώ ότι ο ρόλος που μπορεί να παίξει και οφείλει να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι πάρα πολύ σημαντικός και βεβαίως προσδοκούμε την υλοποίηση του πακέτου των έξι μέτρων και περιμένω φυσικά τις παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Όπως είπα και πριν, κάποιοι θα πρέπει να φύγουν, οπότε θα δεχτούμε τον πρώτο γύρο συντονιστών, ερωτήσεων από τους συντονιστές ή από όσους έχουν ορίσει. Δεν ξέρω ποιος θα κάνει τις ερωτήσεις από το ΕΛΚ. Ξεκινάμε με το Ούντο. Σάρον, ευχαριστώ. Έχουμε γύρω στις 200 ε, ερωτήσεις για τον κύριο Ροστόφσκι και άλλες τόσες για τον ε, κύριο Όλιρεν. Αλλά λόγω του κατεπήγοντος της κατάστασης θα προτιμώ να δώσω τον λόγο στην ε, Άννη Ποδηματά η οποία μόλις ήρθε από την Αθήνα και έχει να κάνει κάποιες ερωτήσεις που θα θέλαμε να ακούσετε. Σας ευχαριστώ πολύ Ούντο, Σάρον, κύριε Επιτροπέ. Όπως ε, ξέρετε, όπως είπατε, χθες το βράδυ είχαμε μια συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων μεταξύ του Πρωθυπουργού του κυρίου Παπανδρέου και του επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης του κυρίου Σαμαρά να σχηματιστεί η κυβέρνηση συνασπισμού με κύριο στόχο την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν ε, από την ελληνική πλευρά βεβαίως, πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν στις 27 ε, Οκτωβρίου και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές. Πρέπει να τα καταφέρουμε, κύριε Επίτροπε, η Κομισιόν και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν τονίσει πολλές φορές στο παρελθόν την ανάγκη εθνικής ενότητας και εθνικής συνεννόησης ως ε, το μοναδικό τρόπο για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ορθή εφαρμογή πολύ δύσκολων μέτρων και πολιτικών. και όπως ξέρετε και τονίσατε πολλές φορές ε, στο παρελθόν ε, ε, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη ακόμα και πριν από την πρόταση για δημοψήφισμα. Οπότε χρειαζόμαστε μια λύση. Έχουμε τώρα μια λύση και κρίσιμο είναι να κοιτάμε προς τα εμπρός και όχι πίσω. Οπότε για να λειτουργήσει η κατάσταση γιατί βεβαίως η κυβέρνηση συνασπισμού είναι ένα μέσο ένα εργαλείο. Για να λειτουργήσει λοιπόν πρέπει να κινητοποιηθεί η κοινωνία. Οπότε η ερώτησή μου προς σας είναι η εξής. Τι μήνυμα μπορείτε να στείλετε στους Έλληνες πολίτες. Μήνυμα το οποίο θα συνεισφέρει σε μια θετική προοπτική γιατί μέχρι τώρα παρόλες τις αδυναμίες, τις λάθος αποφάσεις οι Έλληνες πολίτες συχνά έχουν την αίσθηση πως αποτελούν στόχο και προσβάλλονται και αυτό είναι τελείως αντιπαραγωγικό. Νομίζω πως όλοι πρέπει να αλλάξουμε σελίδα, να κοιτάξουμε προς τα εμπρός. Νομίζω πως η χθες βραδινή απόφαση είναι μια απόφαση κλειδί και νομίζω είμαι πεπισμένη όσον αφορά τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή πως θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να λειτουργήσει. Γιατί είναι προς όφελος της Ελλάδας και της σταθερότητας της Ευρωζώνης συνολικά. Υπάρχει λοιπόν ένα μήνυμα μια θετική προοπτικής από εσάς, από την Κομισιόν. το οποίο θα δώσει μια πίστη στη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας για το τη δύσκολη πορεία που μας περιμένει. Θα ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις ε, λόγω του χρόνου. Σοφή. Ευχαριστώ Σάρων. Ευχαριστώ τον ε, Υπουργό και τον Επίτροπο που ήρθαν, γιατί δεν έκαναν όλη την αντίστοιχη προσπάθεια για να έρθουν εδώ. Θα ήθελα να εκφράσω μια τεράστια ανησυχία και πραγματικά είναι μεγάλη ανησυχία γιατί αν ε, συζητήσετε το θέμα με τους Ευρωπαίους πολίτες, θα διαπιστώσετε σε μέχρι ποιο βαθμό η διαχείριση αυτών των κρίσεων γίνεται αλλού, μακριά από τον πολίτη, σε διαφανείς κύκλους και μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμεύει ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε για τα βιενικά σας λόγια για το εξάπτυχο αυτό πακέτο, αλλά ποια είναι τα αποτελέσματα. Έχω τα συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής Ευρωζώνης και έμεινε εμβρόντιτη από το εξή. Ουδής δεν είχε την επαναστατική ιδέα να περιλάβει στα συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής μερικά από τα στοιχεία που είχαν συζητηθεί στα πλαίσια του εξαπλώφτου πακέτου. Για, για παράδειγμα, το Complier Explain, το Συμβούλιο το είχε φεύγει αυτό την Άνοιξη και καταφέραμε μετά από ολονύκτιες συζητήσεις, όπως θα θυμάστε και οι δύο πολύ καλά, να το δημοσιεύσουμε αυτό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί η peer pressure, η πίεση μεταξύ ομοτήμων δεν μπορεί να γίνεται ε, και κλεισμένο το θυρών, ε, κρυπτό και παραβίστο, αλλά ούτε και αυτό περιλήφθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωζώνης. Κύριε Ροστκόφσκη, εσείς δεν είστε τόσο άμεσα αναμειγμένος, αλλά ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι παιχνίδι παίζετε. Τι παιχνίδι παίζετε. Να υθετούμε κανονισμούς που όλοι χαίρονται και μένουν ενθουσιασμένοι που εγκρίθηκαν και ευχαριστούν το Κοινοβούλιο για τη συνεργασία και δύο εβδομάδες μετά το Συμβούλιο να τα γράφει όλα αυτά στα παλιά του τα παπούσια και ζητώ συγγνώμη για την έκφραση. Πραγματικά αυτό δεν μας δίνει καθόλου, καθόλου εθάριση. δεν, δεν μου αρέσει καθόλου να με κοροϊδεύουν και να με περιγελούν. Γιατί μέσω ημών εμπέζεται και τους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες αυτούς που κάνουν την προσπάθεια και πηγαίνουν και ρίχνουν την ψήφα του στις Και θα ήθελα σήμερα πανηγυρικά, τελετουργικά ενώπιόν σα να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται την κρίση είναι μη δημοκρατικός, απομακρύνει, παραγωνίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι σκαδαλώδη αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης. Κανείς ούτε καν εμεί που για 20 χρόνια της ζωής τους ε, ήταν υπέρ της ε, γαλλογερμανικής συνεργασίας βρίσκονται σε αμηχανία. Δεν μπορούμε να ζητούμε μόνο από δύο πρωτεύουσε να διαχειρίζονται την κρίση. Έχουμε πολύ, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ναι, αλλά απ' την άλλη πώς θέλετε ο ελληνικός λαός να μην αισθάνεται ότι βρίσκεται σε αβάσταχτη κατάσταση. Πώς θέλετε οι Ιταλοί που λαμβάνουν τις τράπεζες τις έκτη, που δεν ξέρουμε ποιος τις έγραψε, πού συζητήθηκαν, λαμβάνουν τις επιστολές από την, από την ΕΚΤ και μάλιστα τις αισθενίζεται και το Συμβούλιο ε, που υιοθετεί πολύ περίεργες καλοπρόσαλες θέσεις στο G20. Πιστεύετε ότι όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα δημοκρατικής και διαφανούς Ευρώπης για τους Ευρωπαίους πολίτες. Όχι και πραγματικά αισθάνομαι ιδιαίτερη ντροπή και ως εισηγήτρια για το εξαπλό αυτό πακέτο των νομοθετικών προτάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το ΕΛΚ μου λέει τώρα ότι θα μιλήσει η Ντανούτα Χιούμπνερ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος από το ΕΛΚ στον κατάλογο μου. Ωραία, οι κυρίες προηγούνται. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα εσείς να απαντήσετε. Βεβαίως υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ε, στον επεκτατικό ρόλο των πακέτων λιτότητας, ότι έτσι αναπτυχθεί η οικονομία. Εγώ δεν συμφωνώ γιατί οι αγορές δεν κοιτάνε μόνο ελλείμματα και χρέη αλλά κοιτάνε και τη δυνατότητα μιας χώρας να επανέλθει στην ανάπτυξη. Οπότε τα πακέτα λιτότητας θα πρέπει να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη. Τέλος πάντων, εγώ δεν πιστεύω σε όλη αυτή την ιστορία. Και τώρα αν δείτε τις αποφάσεις του Οκτωβρίου. Εάν δείτε το 50% αυτή την απομείωση του ελληνικού χρέους για τις ε, για τους ιδιώτες δανειστές. Και αν δείτε δε πως ε, οι τράπεζες μπορούν να φτάσουν το 9% όχι μέσω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αλλά μείωση των ισολογισμών τους, ε, τότε θα δείτε πως θα μειωθούν οι πιθανότητες ανάπτυξης. Μπορούτε λοιπόν, μπορεί να μου πει η Κομισιόν που βλέπει την δυνατότητα του συστήματός μας και της πολιτικής μας να δημιουργήσει ανάπτυξη σε χώρες ε, όπως η Ελλάδα. Και τελευταίος σε αυτό τον γύρο, ο Φιλίπ. Ευχαριστώ, θα μιλήσω αγγλικά. Κύριε Πετροπέ, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που ήρθατε, ειδικά σήμερα. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είναι στη μελέτη μας, θα πω μόνο ένα πράγμα. Χρειαζόμαστε μια πιο συνολική, ολοκληρωμένη οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Αυτό είναι σαφές και το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι απολύτως απαραίτητο όσον αφορά τη διαδικασία. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε πως πρώτον θα λειτουργεί σύνεπως και όλες οι μελέτες έχουν δείξει πως έχουμε κάποια προβλήματα όσον αφορά την πολιτική συνέπεια μεταξύ των, χωρών, των συστάσεων χωρών και όσον αφορά τη στρατηγική 2020 κτλ. Δεν θα επεκταθώ για μένα. Το βασικό είναι η στήριξη του λαού. Γνωρίζουμε πως οι πολιτικές που επιβάλλονται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη ως μέρος ε, της επίγουσας βοήθειας και της οικονομικής αυτής διοίκησης δεν έχουν τη στήριξη του λαού. Και μπορεί να ασκεί κανεί κριτική στην υπόθεση αυτή του δημοψηφίσματο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μα στηρίξει ο λαό. Εκεί που βλέπω εγώ το μεγαλύτερο κίνδυνο στο εξάμεινο αυτό είναι στην έλλειψη δημοκρατική λογοδοσία. Και ε, ασκώ κριτική και στο Κοινοβούλιο αυτό όταν θέλει να διαχειρίζεται κάθε βήμα κάθε θεσμικής ε, διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. είναι αυτό ο ρόλος μας. Αντιθέτως, σε σημεία κλειδιά των αποφάσεων, όταν κατευθύνουμε οικονομικέ, πολιτικέ, δημοσιονομικέ στρατηγικέ, και οι προσανατολισμοί αυτοί θα γίνουν και πιο υποχρεωτικοί και δεσμευτικοί, νομίζω πως σε κρίσιμες στιγμές θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατική στήριξη και με αυτό εννοώ στήριξη και ε, ψήφιση τουλάχιστον από αυτό το κοινοβούλιο. Δεν θέλω να να ζητήσω εξουσίες περισσότερες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά όταν κάνετε αυτή την έρευνα της ετήσιας ανάπτυξης που ουσιαστικά είναι κατευθυντήριες, οικονομικές κατευθυντήριες γραμμές και έτσι πρέπει να τις λέμε, αυτό είναι και χρειάζονται. Πρέπει να υπάρχει σε αυτό συναπόφαση. Και αν είναι να είμαστε γρήγοροι, να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε γρήγοροι. Αλλά αυτές είναι χαρακτηριστικές στιγμές όπου πρέπει να διευρυνθεί η πολιτική στήριξη. Αλλιώς ανησυχώ για το ότι η κοινή οικονομική διακυβέρνηση, η ολοκληρωμένη αυτή η οικονομική διακυβέρνηση που χρειαζόμαστε θα σκοντάψει στην έλλειψη πολιτικής στήριξης και μετά θα οδηγηθεί η Ευρώπη σε πολιτική διάλυση, κάτι το οποίο κανείς μας δεν νομίζω ότι θέλει. Οπότε σας παρακαλώ να ξαναδείτε τη διαδικασία για να έχουμε περισσότερη δημοκρατική λογοδοσία. Και εννοώ στην στρατηγική 2020 που είναι δεσμευτική και στην απόφαση και στην ετήσια αυτή μελέτη της ανάπτυξης. Για να στείλουμε ένα μήνυμα στους πολίτες μας πως πράγματι δεν θα αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κλεισμένων των θυρών. Συχνά λέμε πως το Συμβούλιο λειτουργεί και κλεισμένο των θυρών. Ε, ας πούμε πως ε, και η δουλειά της Τρόικας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες είναι ακριβώς αυτό. Δουλεύουν και κλεισμένων των θυρών νομίζω πως σε κάποια κρίσιμα σημεία πρέπει να μπορούμε να πάμε στον Ευρωπαίο πολίτη να του πούμε πως, να του πούμε πως υπάρχει στήριξη. Γιατί δεν αποφασίζει όλη η ΡΕΝ, η Κομισιόν, η Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε τη στήριξη του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Απαντήσεις ε, θα πάρουμε τώρα. Κύριε Υπουργέ, εσείς που πρέπει να φύγετε, θέλετε να μιλήσετε πρώτος, να απαντήσετε πρώτος παρατηρήσει εκτός μικροφώνου, δεν τις ακούμε. Ναι, μου είχε πει ότι θα φύγει ε, τις ε, παρατέταρτο. Τέσσερις παρατέταρτο. Και θα τον αντικαταστήσει, θα έρθει ένας γενικός γραμματέας. Okay. A θέλετε να θέσετε το ερώτημά σας, αλλά μήπως δεν απαντηθεί. Εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πολύ, Σάρων. Όπως ε, μια και διάφοροι σκιώδεις εισηγητές ε, παρενέβησαν. Νομίζω ότι θα μπορούσα και εγώ να μιλήσω άμεσα με τον κύριο Επίτροπο και τον ε, κύριο Υπουργό. Θα πάω όμως απευθείας ε, στα πιο σημαντικά ζητήματα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, αυτό το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έτσι όπως έχει μπει στο τραπέζι φαίνεται σαν μια καθαρά γραφειοκρατική άσκηση. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε από τη στιγμή που ε, βρεθήκαμε με το ευρώ είναι να δημιουργήσουμε ένα καλό σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης ε, και βεβαίως αυτή η οικονομική διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει μέσα από τη γραφειοκρατία και μόνο. Και νομίζω ότι σήμερα όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται ε, για τη δημοκρατική λογοδοσία είναι ότι στην ουσία η λογοδοσία αυτή δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να κάνουμε ευρωπαϊκό εξάμεινο, δεν μπορούμε ε, να βρισκόμαστε στο τιμόνι μιας οικονομικής ευρωπαϊκής διακυβέρνησης χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία. Σε ένα εθνικό κοινοβούλιο τα πράγματα είναι απλά. Γιατί έχουμε ε, τους, ε, τους, ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Ε, έχουμε ας πούμε και αυτό που είπε, εδώ έχουμε αυτό που είπε ε, ο Στέλφος Λαμπέρ, ε, δηλαδή έχουμε κάποιες οικονομικές προοπτικές οι οποίες μας οδηγούν. Όμως θα πρέπει να περάσουμε σε μια κατάσταση όπου το κεντρικό σημείο αναφοράς θα είναι το, το Europlus και τότε θα έχουμε διπλή δημοκρατική άρνηση Απ' τη μία το κοινοβούλιο δεν θα μπορεί να κάνει κάτι και απ' την άλλη εσείς θα μας λέτε ότι, ε, ότι εσείς δημιουργείτε έχοντας σαν βάση ένα εργαλείο ενώ στο Συμβούλιο η βάση θα είναι διαφορετική και τα εργαλεία θα είναι διαφορετικά. Ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι ε, αγορητές οι οποίοι έχουν εγγραφεί αλλά θα πρέπει να απαντήσει ο κ. Ζωτόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση δεν ε, άκουσα μέχρι τώρα καμία αναφορά στο Europlus, στο Συμβούλιο. Ενδεχομένως αυτό που λέτε να ισχύσει στο μέλλον, αλλά δεν το γνωρίζω και δεν έχει συζητηθεί. Δεν ε, ξέρω, τουλάχιστον δεν γνωρίζω, κανένα τέτοιο διαβολικό σχέδιο. Πρέπει να πω ότι και σαν Πολωνική Προεδρία και εγώ ο ίδιος προσωπικά ε, πιστεύουμε ότι και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να ασχολούνται περισσότερο, να έχουν μεγαλύτερο λόγο για τα οικονομικά. Ε, αυτή είναι η θέση μας. Και είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες εθνικές κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες επιβεβαιώνει ε, η Κομισιόν και τις οποίες ε, γνωρίζει ε, μονάχα αφότου, αφότου οι εθνικές κυβερνήσεις τις κυκλοφορήσουν και είναι θεμητό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να ελέγχει αυτές τις προοπτικές. Τώρα, Ετέθη και ένα ερώτημα σχετικά με τις πολιτικές σύγκλησης κλπ. Στην ουσία αυτό το οποίο συζητάμε εδώ έχω την αίσθηση ε, ότι είναι το εξής. Stable public finances. Um, Εάν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μια σταθερή οικονομική κατάσταση, θα πρέπει να έχουμε σαφή πολιτική διαρθρωτικών πολιτικών που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Και κατά αυτήν την έννοια πιστεύω ότι πολύ χρήσιμο θα ήταν να ενισχυθούν αυτές οι συστάσεις και να ενισχυθεί βεβαίως ε, και η δημοκρατική λογοδοσία και το περιεχόμενο της δημοκρατικής εντολής. Βεβαίως, ε, δημοκρατική λογοδοσία και δημοκρατική εντολή μπορεί να περιέχουν πολλά πράγματα, αλλά εγώ είμαι υπέρ και των δύο. Και απαντώ σε τρία ερωτήματα που είχαν αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά ε, το ζήτημα που έθιξε η κυρία Χιούμπνερ, ε, στα περάσματα ΕΚΟΦΗΝΕ αναφέρεται σαφώς ότι το EPA θα πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο ώστε ε, η νέα κεφαλιακή επάρκεια ε, και η απέτηση του 9% ε, να μην αφορά τα ισοζύγια, αλλά βεβαίως είναι σαφές ότι το πράγμα δεν είναι καθόλου εύκολο. Και φυσικά θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί όσον αφορά όλα αυτά τα ζητήματα που έχει θίξει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ε, έχει δίκιο η κυρία Χιούμπνερ ε, όταν λέει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ότι εάν όλες οι χώρες προσπαθήσουν να εξηγιάνουν τα δημοσιονομικά τους, σαφώς ε, δεν θα οδηγηθούμε σε ανάπτυξη. Υπάρχουν και χώρες όμως οι οποίες έχουν ισχυρή δημοσιονομική θέση και οι οποίες ε, προσπαθούν να πάρουν αντισταθμιστικά μέτρα, να κάνουν αντισταθμιστικές ε, ε, κινήσεις. Αλλά είναι λίγες αυτές οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. και η κλασική κινσιανή πολιτική που έχει ακολουθηθεί οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μια τέτοια κίνηση από πλευράς τραπεζών τελικά θα αντιτίθεται στις συνθήκες. Νομίζω ότι με αυτά απήντησα στις ερωτήσεις. Όλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σάρων. Θα ξεκινήσω με την ερώτηση και σχόλιο της κυρίας Πόδηματά όσον αφορά την Ελλάδα. Είναι σαφές πως η Ευρώπη είναι στο πλευρό της Ελλάδας. Είμαστε εταίροι της Ελλάδας και των Ελλήνων πολιτών για να ξεπεράσουν την σοβαρή αυτή κρίση που είναι αποτέλεσμα λαθών του παρελθόντος στην δημοσιονομική και οικονομική πολιτική. Βεβαίως είναι μια σχέση αμφιδρομή. Μπορούμε να το περιγράψουμε ως ένα είδος ε, κοινωνικού συμβολέου μεταξύ της Ελλάδας και της υπόλοιπης Ευρωζώνης υπό την έννοια πως η Ευρωζώνη συμφώνησε να στηρίξει την Ελλάδα υπό τον όρο πως η Ελλάδα θα σταματήσει να ζει πέρα από τις δυνατότητες της και θα αποκαταστήσει την οικονομική ισορροπία, το οποίο σημαίνει πως αναμένουμε πως η Ελλάδα θα εκπληρώσει τις δεσμές που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος της Ένωσης και του Δονοτού και της τελευταίας συνόδου της 27 Οκτωβρίου. Και γι' αυτό, όπως είπατε κι εσείς, έχει πράγματι μεγάλη σημασία να έχουμε ευρύτερη εθνική ενότητα και τώρα είμαστε στην διαδικασία αυτή και αναμένω πως ε, θα υπάρξει μια συμμαχική κυβέρνηση εθνικής ενότητας σύντομα στην Ελλάδα και για το όφελος ε, των Ελλήνων πολιτών. Και βεβαίως οι πτυχές ε, της ανάπτυξης και της μεταρρύθμισης είναι σημαντικές. Δεν έχει μόνο σημασία η δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά και η στήριξη της ανάπτυξης στην Ελλάδα. Γι' αυτό η ομάδα δράσης που έχουμε συστήσει εργάζεται με σκοπό να διευκολύνει μια γρηγορότερη και καλύτερη απορρόφηση των ε, κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων για να αυξηθούν οι επενδύσεις και οι θέσεις εργασίας και να δώσει τεχνική αρρωγή σε κάποιους ε, κέριους τομείς, ε, είτε μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε για την φορολογία, όπου σαφώς χρειάζεται με βάση τις πρόσφατες εμπειρίες. Οπότε, σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα υποστηρίζουμε την Ελλάδα και αναμένουμε πως η Ελλάδα από την πλευρά της θα τηρήσει τη συμφωνία. Όσον αφορά αυτά τα οποία είπε η Ντανίτα Χιμπνερ και η κυρία Ποδηματά, όσον αφορά δηλαδή την ανάπτυξη, πέρα από τα ζητήματα του πώς η ομάδα δράσης στηρίζει την ανάπτυξη και βεβαίως δεν είναι μόνο η δική της Κομισιόν αλλά και των κρατών μελών γιατί έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από την Κομισιόν σε κάποιους τομείς βλέπουμε πως ε, μια κλασική και ενσιανή πολιτική σε μια κατάσταση στην οποία τα επίπεδα του χρέους ε, φτάνουν ε, 80-90% του ΕΠ δεν είναι ο κατάλληλος δρόμος. Ανταυτού, ε, κατ' ουσίαν μιλάμε για μηδενική ανάπτυξη προς το τέλος του έτους ε, και αυτό έχει σχέση με την έλλειψη εμπιστοσύνης στην οικονομία και ορισμένες φορές ε, στην διαμόρφωση της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, κατά την άποψή μου, το κλειδί για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη είναι να λυθεί η κρίση του δημοσίου χρέους και να περιορίσουμε τον αντίκτυπό της στον τραπεζικό τομέα και να διασφαλίσουμε έτσι πως η πίστη η οποία θα διατίθεται στους πολίτες μας και στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά θα παραμείνει η ίδια και άρα θα καθυσυχαστούν αυτοί. Γιατί, Γιατί οι αναταραχές αυτή τη στιγμή της ε, αγοράς ε, διαβρώνουν τα θεμέλια της οικονομίας και της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Πρέπει πρώτα απ' όλα λοιπόν να, σταματήσει, να σταματήσουν αυτές οι αναταραχές στην αγορά και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πιστικά μέτρα και στον τομέα της κρίσης του δημοσίου χρέους και με την διασφάλιση επαρκούς ε, βαρότητα στον τραπεζικό τομέα. Όσον αφορά αυτά τα οποία είπε η κυρία Γκουλάντ για την σύνοδο κορυφής της Ευρωζώνης και κάποια συμπεράσματα τα οποία συμπίπτουν. Έχετε δίκιο όπως λένε και στα λατινικά, αν δεν κάνω λάθος, η επανάληψη είναι μήτρη της μαθήσεως. Οπότε δεν βλάπτει. Εάν στα συμπεράσματα ε, επαναλαμβάνουμε κάποια πράγματα, στα συμπεράσματα της Ευρωζώνης, ε, ε, κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν στο πακέτο των έξι οδηγιών. Παραδείγματο χάρη ε, οι κανόνε για ισοσκελισμένου προπολογισμού, οδηγία για τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια, πρόσκληση στα εθνικά κοινοβούλια να σεβαστούν τι ε, συστάσει οικονομική και δημοσιονομική πολιτική είναι σημαντικά και ελπίζω να, το, να συμφωνήσετε κι εσείς, δέσμευση να συμφωνήσουμε με τις συστάσεις της ε, Κομισιόν όσον αφορά το σεβασμό του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Ορίστε. Αν μου επιτρέπετε, δεν είναι καν επανάληψη. Είναι παράληψη. Παρέλειψαν να συμπεράβουν τη δική μας προσθήκη στο εξαπλό αυτό πακέτο. Και να μας εξηγήσετε ότι αυτό που διαγράψατε από τα συμπεράσματα είναι αυτό ακριβώς που ε, προτείναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω ήταν τυχαίο. Δεν με ε, εμένα καθόλου δεν με συμφέρει αυτή η διαγραφή. Το αντίθετο. Εγώ θα ήθελα οι υπουργοί και οι υφυπουργοί πραγματικά να έρθουν και να δώσουν λόγο εκ μέρους, της, εκ των κυβερνήσεών τους σε ό,τι αφορά τις ε, οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές. Μα ακριβώς γι' αυτό το λόγο το επισήμανα και δημοσίως, ε, κύριε Επιτροπέ. Νομίζω ότι συμφωνούμε και ως προς το σημείο αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, δημοκρατική λογοδοσία και την Ευρώπη μετά την εφαρμογή των εξ αυτών οδηγιών. Η κυρία Μπέρες μίλησε για την σημασία που έχει η δημοκρατική λογοδοσία στα πλαίσια του εξαπλού αυτού πακέτου. Το άκουσα και στο Συμβούλιο και στις διασκέψεις κορυφής αυτό το θέμα πολλές φορές, αλλά σας διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συμπεριλάβει ε, το πακέτο Ευρωπλάς ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και στο πακέτο της δημοσιονομικής ε, εποπτείας. Και θέλουμε να το κάνουμε αυτό στα πλαίσια της ετήσιας ε, επισκόπησης που θα υποβάλουμε το αργότερο τέλη Νοεμβρίου και στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και στο ίδιο αυτό πλαίσιο προτιθέμεθα να υποβάλουμε και την πρότασή μας για τα μελλοντικά βήματα προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση και κατά πάσα πιθανότητα θα δημοσιεύσουμε και το, την πράσινη βίβλο για την σταθερότητα του ευρώ. Και μέσω και με βράχη μέσω πρόθεσμα υπάρχουν τέτοιε προτάσει και για φόρα ανάπτυξη και για δημιουργία θέσεων απασχόληση. Τώρα, πολύ ευχαρίστω να επανέλθω στι 23 Νοεμβρίου στην Επιτροπή σα μετά την παρουσίαση και του, ε, της αιτήσιας επισκόπησης και των ε, συμπληρωματικών προτάσεων για την ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση, καθώς και την πράσινη βίβλο για τη σταθερότητα. Ε, από ό,τι φαίνεται σε λίγο θα φύγει και ο Επίτροπος. Κύριε Χουντή, ε, θα σας δώσω το λόγο για να υποβάλλετε δική σας ερώτηση και μετά ίσως εκτός μικρόφωνου. Ο κύριος Χουντής είχε ζητήσει το λόγο πολύ πριν από εσάς, κύριε μου. Ε, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε έτσι όπως εξελίχθηκε η διαδικασία δεν έχω τη δυνατότητα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και επομένως θα απευθυνθώ στον κύριο Ρεν, ειλικρινά τον ευχαριστώ, διότι, ναι, διότι κατά τη διάρκεια των απαντήσεων και των δευτερολογιών προσπάθησε να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις που γραπτά είχαμε υποβάλει σε σχέση με το εξάμεινο. Όμως, με βάση τη συγκυρία, κύριε Ρεν, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν δημοσιεύματα στον τύπο ότι υπάρχει έκθεση της νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που μελετάει σενάρια για πιθανότητα εξόδου μιας χώρας από την ζώνη του ευρώ. Αυτό, όπως γνωρίζουμε, δεν προβλέπεται από τις συνθήκες. Άρα έχουμε καινούργιε ερμηνείε. Ταυτοχρόνως, το Σαββατοκύριακο κάνετε μια δήλωση ότι δεν θέλουμε την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε περίπτωση και για αυτό το ενδεχόμενο. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, υπάρχει τέτοια έκθεση κύριε Επίτροπε. Δεύτερο, τι προβλέπουν τα σενάρια της έκθεσης σε σχέση με τη συνθήκη. Και τρίτο, γιατί όχι, θα πάρουμε εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια τέτοια έκθεση να ξέρουμε τι προβλέπετε, τι προετοιμασία γίνεται. Πιστεύω ότι αυτά που είπατε δεν τα είπατε χωρίς να έχετε κάτι στο νου, παρά το γεγονός ότι ξαναλέω μια τέτοια περίπτωση δεν προβλέπεται από τη συνθήκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. no such study to which... ευχαριστώ δεν υπάρχει αυτή η μελέτη στην οποία αναφερθήκατε. Βεβαίως η Κομισιόν, όπως κάθε οργανισμός που έχει ευθύνες για το μέλλον και την ευημερία της Ευρώπης και των Ευρωπαίων πολιτών, πρέπει να καταρτίζει κάποια σενάρια και να είμαστε προετοιμασμένοι για διάφορα σενάρια. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια μελέτη σαν αυτή που αναφέρατε. Τώρα στην Ελλάδα ε, έχει ουσιαστική σημασία οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας να μπορέσουν να διαλέξουν την ενότητα και να θέσουν σε πρώτη μοίρα την ευημερία των πολιτών τους. Και ελπίζω να οδηγηθούμε τώρα σε μια συμμαχική κυβέρνηση εθνικής ενότητας και αυτά τα αρνητικά σενάρια να μην χρειαστεί να τα σκεφτούμε και να διασφαλίσουμε από κοινού πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι μέλος Ευρωζώνης που είναι η θέση της Κομισιόν. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ε, η Ελλάδα να μπορεί και να παραμείνει ε, στην Ευρωζώνη. Και είμαστε οπισμένοι πως η Ελλάδα θα πείσει τους εταίρους της πως θα μπορέσει να κάνει αυτό που της αναλογεί με αυτή τη συμφωνία. Ήρθε η σειρά σου. Ευχαριστώ. Νόμιζα ότι ε, προσπαθούσαμε να αποκαταστήσουμε μια ισορροπία μεταξύ μικρών και μεγάλων χωρών, μικρών και μεγάλων ομάδων. Αυτό φανταζόμουν και στη συζήτηση. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, ιδιαίτερα για τη σημασία της ανάκτησης της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των καταναλωτών και φυσικά και την λαϊκή υποστήριξη. Είναι αλληλένδετα όλα αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα ε, δημοκρατικής ε, λογοδοσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερο μας ενδιαφέρει αυτή η δημοκρατική λογοδοσία των, των κρατών μελών, των κυβερνήσεων απέναντι στο λαό. Είχαμε πολλές αναταραχές την προηγούμενη εβδομάδα και ζητούμε περισσότερο κάποιες οδηγίες από σας, κάποιες ε, καταθεντήρες γραμμές. Πιστεύετε ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο λειτουργεί διαφορετικά για τις ζώνες εντός και εκτός ευρωζώνης και ιδιαίτερα για τις χώρες που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να ενταχθούν στο ευρώ αλλά δεν έχουν ε, μπει ακόμη στην ευρωζώνη. Μετά τις συζητήσεις των τελευταίων εβδομάδων, χρήσιμο θα ήταν κύριε Επίτροπε να μας πείτε τη γνώμη σας και για τις χώρες που έχουν αναλάβει τη δέσμευση αλλά δεν έχουν ακόμη ε, μπει στο ευρώ. Γιατί τουλάχιστον μία από τις χώρες αυτές ε, ίσως θα ήθελε ε, να απευθυνθεί στο λαό και να εξασφαλίσει την λαϊκή υποστήριξη για την είσοδο στο ευρώ. Πώς επηρεάζει λοιπόν το ευρωπαϊκό εξάμεινο τι χώρε εντό και εκτό ευρώ, αυτέ που έχουν δεσμευτεί και αυτέ που δεν έχουν καν δεσμευτεί, ώστε να εξασφαλίσουμε πραγματικά και για τι χώρε αυτέ τη λαϊκή υποστήριξη για την προσχώρηση στην Ευρωζώνη και το ευρώ. Ευχαριστώ. Είναι φυσικά σημαντικό να κερδίσουμε την υποστήριξη του κόσμου για τις μεταρρυθμίσεις που συμφωνήσαμε. Και πραγματικά προσβλέπω σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με τα Εθνικά Κοινοβούλια γιατί νομίζω ότι είναι κοινό αυτό το καθήκον να αναμίξουμε και τα εθνικά κοινοβούλια για να έχουν και αυτά την αίσθηση ότι συμμετέχουν στη νέα εργαλειοθήκη, στον αυτό το μηχανισμό, το πακέτο των έξι ε, οδηγιών, γιατί νομίζω ότι με το πακέτο αυτό εξυπηρετούνται και οι στόχοι και των εθνικών κοινοβουλίων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας για τις διαφορές ε, εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στις χώρες εντός και εκτός της Ευρωζώνης. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν προϋποθέτει διακρίσεις μεταξύ Ευρωζώνης και χωρών εκτός Ευρωζώνης. Υπάρχουν ενηλογικές διαφορές και οι χώρες της ε, Ευρωζώνης υποβάλλουν προγράμματα σταθερότητας, ενώ οι υπόλοιπες χώρες εκτός Ευρωζώνης υποβάλλουν προγράμματα σύγκλησης οι διαφορέ όμω μεταξύ προγραμμάτων σταθερότητα και προγραμμάτων σύγκληση είναι απειροελάχιστε. Τώρα, οι διατάξει ε, του εξαπλού πακέτου εφαρμόζονται μόνο στι χώρε Ευρωζώνη και άρα δεν εμπίπτουν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Βέβαια, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δημιουργεί ένα πλαίσιο για τα νέα εργαλεία, τους νέους μηχανισμούς του εξαπλού πακέτου και για την εφαρμογή τους. Οπότε από αυτή την άποψη η διαφορά αφορά περισσότερο τη δέσμευση για βαθύτερη οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση και όλο και πιο στενή οικονομική ένωση. Ενώ η συμμετοχή στην Ευρω... Ε, από τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη. Και κατά κάποιο τρόπο η δέσμευση προϋποθέτει και την ε, προθυμία ενίσχυσης, ε, ενισχυμένης εφαρμογής των κανόνων που εφαρμόζονται στην Ευρωζώνη και περιλαμβάνονται στο εξαπλό πακέτο. Οπότε αυτή την άποψη το ευρωπαϊκό εξάμεινο ε, ισχύει για όλες τις χώρες μέλη για τις 27 δηλαδή. Σας ευχαριστώ για τα πολύ εύστοχες οι ερωτήσεις σας, πολύ μεστές. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά είχα ανηλυμένη υποχρέωση. Σε λίγο θα αρχίσει και η συνεδρίαση του Eurogroup, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να παραστώ. Η διαχείριση το, της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο σημαντικότερο σημείο, γι' αυτό θα πρέπει να φύγω να πω στο Συμβούλιο, αλλά θα τα πούμε και πάλι σύντομα για την ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση και την ε, ε, έκθεση της επισκόπησης. Τρεις ακόμη ομιλητές εκδήλωσαν την επιθυμία να υποβάλουν ε, ερωτήσεις. Έχουμε όμως τον Υφυπουργό που θα εκπροσωπήσει εδώ την Πολωνική Προεδρία και θα απαντήσει ερωτήσεις. Πάντως στόχος της ακρόασης ήταν να διερευνήσουμε το γιατί στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ορισμένες προτάσεις της Επιτροπής αλλοιώθηκαν κάπως και αμβλήθηκαν. Λυπάμαι Σάρων, αλλά είχα ερώτηση προς τον Επίτροπο που έφυγε. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Η κρίση συνεχίζεται και πρέπει να τη χειριστούμε. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας, έχω και εγώ μια ερώτηση. Κατά την άποψή μου η σύνοδος κορυφής των G20 Σκάνες ήταν μεγάλη απογοητεύση. Χάσαμε μία ευκαιρία αντί να στείλουμε ένα μήνυμα εμπιστοσύνης που θα καθησύχαζε τον κόσμο δείξαμε πως δεν πιστεύουμε και οι ίδιοι σε αυτά τα οποία λέμε. Ήταν η Ιωνή κακή, ο καιρός ήταν άσχημος, το δημοψήφισμα από την Ελλάδα αποτελούσε έκπληξη και δεν υπήρχε και πάρα πολλής χρόνος για να συζητούν τα ανοιχτά ζητήματα. Τι συνέβη λοιπόν. Πρώτα αυτό το οποίο ήταν εδώ και καιρό ταμπού, δηλαδή η εγκατάλειψη μιας χώρας, μιας, της Ευρωζώνης από μια χώρα. Αυτό λοιπόν το οποίο ήταν εδώ και καιρό ταμπού να φύγει μια χώρα από την Ευρωζώνη, ξαφνικά θεωρείται μια ρεαλιστική πιθανότητα. Αυτό ήταν άσχημο μήνυμα. Το δεύτερο ξεκινήσαμε να συζητάμε μήπως πέρα από τη μόχλευση του ΙΕΦΣΕΦ ε, χρειάζονται και άλλα μέτρα όπως ε, παραδείγματος χάρη να χρησιμοποιηθούν τα νομισματικά αποθέματα ακόμα και τα αποθέματα χρυσού για να δοθεί μεγαλύτερη πυρή, ε, πυρός στο EFSF. Αυτό δείχνει στους πολίτες και στις αγορές πως δεν πιστεύουμε και οι ίδιοι πως επαρκεί αυτό το οποίο αποφασίσαμε πριν από λίγες εβδομάδες και έτσι δεν καθυσυχάζουμε. Δεύτερον, δεν στείλαμε ένα σαφές μήνυμα πως οι παγκόσμιες δυνάμεις, οι G20 δηλαδή, πραγματικά συμφωνούν όλοι. Ο καθένας προσπάθησε να δώσει συμβουλές στον άλλον και οι ΗΠΑ δεν νομίζω να βρισκόνται σε πολύ καλύτερη θέση από την Ευρώπη. Ήδη σήμερα άκουσα πως οι Κινέζοι έχουν τον κίνδυνο κόμμα 3 εκατομμυρίων σε ε, δάνεια μέσω, ήδη, μέσω ιδιωτικών τραπεζών και βεβαίως από την άλλη υπάρχει και η Ελλάδα και κάποιοι στους ε, G20 ξεκαθάρισαν, δεν θέλω τώρα να τους πω, πως δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα στην συμπεριφορά τους. Όλα αυτά κατά την άποψή μου, περισσότερο τρόμαξαν παρά καθυσίχασαν και έστειλαν θετικό μήνυμα στις αγορές. Και αναρωτιέμαι αν είναι πραγματικά απαραίτητο να αποφεύγουμε τέτοια πράγματα. Thank you for... Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Όμως ως Προεδρία δεν ε, ήμασταν στην διάσκεψη των κανόν γιατί αυτό είναι προνόμιο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπότε η Πολωνική Προεδρία δεν ήταν παρούσα. Σε κάποιο βαθμό βεβαίως συμφωνώ με την άποψή σας. για την κατάσταση στις ε, Κάνες. Υπάρχει λοιπόν ακόμα έλλειψη πολιτικής συμφωνίας για τα μέτρα τα οποία χρειάζονται σε αυτή την σοβαρή κατάσταση, αλλά νομίζω πως δεν είναι η τελευταία φετινή συνάντηση. Νομίζω πως μπορούμε να αναμένουμε και άλλες ε, συναντήσεις των φόρων αυτών για να συζητήσουμε περισσότερο και πιθανώς να λύσουμε, να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες θα συζητήσουμε την συνάντηση των G20 και την συνέχεια των συνόδων κορυφής της Ευρωζώνης αύριο στο Συμβούλιο Εκοφήν και βεβαίως νομίζω πως κάποια ζητήματα από αυτά που ετέθησαν εδώ σήμερα στο Κοινοβούλιο θα συζητηθούν πιο λεπτομερώς. Οπότε νομίζω πως θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες ε, λύσεις. Όμως αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να απαντήσω ή ικανοποιητικά. Ευχαριστώ. Ούντο. Ναι. Καλό είναι το ότι ήρθε ο κύριος Υφυπουργός για να συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά. Θεωρώ πως ένα ζήτημα της ε, συναδέλφου Χίμπνερ δεν έχει απαντηθεί, δηλαδή το πώς θα προχωρήσει η δύσκολη διαδικασία της ανάπτυξης και ε, δικαίως είπε πως δεν θα προκύψει ανάπτυξη μόνο από τη λιτότητα και ακούσαμε τον πρόεδρο του Συμβουλίου και την Κομισιόν πως δεν ε, εμπιστεύονται ενσιανά μέτρα, αλλά πρέπει να λυθεί η λύση του δημοσίου χρέους. Έχω ερώτημα τώρα προς την Προεδρία του Συμβουλίου, γιατί ξέρω πως και εσείς κύριε Υφυπουργέ πάντα ήσασταν υπέρ της ε, νομοθεσίας για τις χρηματαγορές. Ανάπτυξη, λέει η Κομισιόν ε, και η Προεδρία του Συμβουλίου, δεν μπορούμε να την προωθήσουμε την ανάπτυξη γιατί πρέπει να λυθεί η κρίση του δημοσίου χρέους όταν κάνουμε εμεί εδώ μέσα νομοθεσία, όπως ε, παραδείγματο χάρη ο κύριος Γκέιμπελς, ο κύριος Κοφάν και άλλοι. Ε, χρειαζόμαστε πάνω από ένα χρόνο για να ρυθμίσουμε τα μέσα τα οποία είναι υπεύθυνα από ό,τι φαίνεται για την κλιμάκωση της ε, κρίσης του δημοσίου χρέους του καλοκαίρι στην Ιταλία. Μιλάω για το credit default swaps και βεβαίως ε, μας μπλοκάρει το Συμβούλιο και μας λέει πως δεν χρειάζεται να οργανώσουμε την ανάπτυξη ανταυτού να λύσουμε την ε, χρήση του δημοσίου χρέους. Έχουμε μεγάλες αντιπαραθέσεις που έγιναν εδώ πέρα για τα hedge funds, τις κοιόδεις τράπεζες και λέμε πως δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά. Μας μπλοκάρει ξανά το Συμβούλιο και πάμε τώρα και ακούμε στους G20 πως ξαφνικά προκύπτει μία έκπληξη πως είναι πρόβλημα αυτές οι σκιώδεις τράπεζες που δεν το ξέραμε. Μέχρι πότε και ε, δεν ε, απευθύνομαι σε σας προσωπικά γιατί ξέρω πως εσείς πραγματικά το θέλετε αυτό. Εννοώ το Συμβούλιο όμως. Πόσο, το, πόσο καιρό το Συμβούλιο θα κρατάει στο σκοτάδι το την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη όσον αφορά τα στοιχεία της κρίσης. Είναι βασικό πρόβλημα της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν ονομάζουμε καν το ποιος εδώ πέρα μπλοκάρει και σταματάει την νομοθεσία για τις ε, χρηματαγορές. Είναι αυτή η κατάσταση απαράδεκτη γιατί το πρόβλημα συνεχώς αναβάλλεται χωρίς να λύνεται και Κανείς φταίει, κανείς δεν είναι υπεύθυνο και κανείς δεν έκανε τίποτα. Εδώ πέρα υπάρχει βασικό δημοκρατικό κενό και δεν βρίσκεται στο κοινοβούλιο. Είναι στο συμβούλιο. Γιατί λένε άλλα πράγματα στις χώρες τους από αυτά που κάνουν στις Βρυξέλλες. Και το ίδιο ισχύει και για το πακέτο οικονομικής ε, διακυβέρνησης όπου θα έχουμε αφενός τρία είδη δικαίου. Έχουμε το εξαπλό πακέτο, έχουμε το σύμφωνο του ευρώ συν, το οποίο δεν πέρασε ποτέ από το κοινοβούλιο με τη συναπόφαση και έχουμε παλαιές θέσεις όπως παραδείγματο χάρη την διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις καθητήρες γραμμή για την απασχόληση που προφανώς δεν παίζουν κανένα ρόλο πλέον. Όλα αυτά είναι ευθύνη και συνυπευθυνότητα σε άλλες περιπτώσεις του Συμβουλίου, είναι αδιαφανή και συνεισφέρουν σε αυτή την κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε κάποια στιγμή ποιο φέρει την ευθύνη για το κάθε πράγμα. Thank Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω από το Ευρωπαϊκό Εξάμενο, που είναι και το κύριο θέμα αυτής της ακρόασης και της συζήτησης. Δεν θα ήθελα στο στάδιο αυτό να τροποποιήσουμε το σύστημα χωρίς ακόμη να έχουμε κάνει αξιολόγηση, χωρίς καν να έχουμε ε, δει πώς λειτουργεί αυτό το εξάμεινο πειραματικά. Γιατί είναι η πρώτη περίοδος εφαρμογής του. Του χρόνου θα έχουμε την ευκαιρία και νομίζω θα είναι πιο σκόπιμο να εξετάσουμε και το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τη στάση του και, και το θέμα της διαφάνειας που επισημάνατε. Αλλά του χρόνου, όχι από τώρα. Ήδη σήμερα όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε αυτό το θέμα να το συμπεριλάβει στο πρόγραμμα εργασιών για του χρόνου. Πάντως, επαναλαμβάνω, είναι πολύ πρόημο να αξιολογήσουμε από τώρα με ποιο τρόπο και σε τι βάση θα κάνει την αξιολόγηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προβήσει στις στάσεις της. Πρέπει πρώτα να δούμε πώς λειτουργεί το εξάμεινο, αν είναι αποτελεσματικό και μετά, μετά από αυτή την αξιολόγηση να δούμε αν την αλλάξει. Πάντως, για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, τα μόνα διδάγματα που μπορούμε να αντιλήσουμε προς το παρόν είναι τεχνικής φύσης. Καλύτερα να αφήσουμε προς το παρόν κατά μέρος την εξαγωγή συμπερασμάτων. Βέβαια, πολύ σωστά επισημάνατε το διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων και εντατικοποίηση αυτού του διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων, ιδιαίτερα για τις οικονομικές πολιτικές και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, γιατί το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα προσφέρει το πλαίσιο για τις συζητήσεις αυτές. Στο εξαπλώ αυτό πακέτο στις έξι νομοθετικές προτάσεις συμφωνήσαμε για αυτό τον οικονομικό διάλογο και θέσαμε τα θεμέλια αυτού του οικονομικού διαλόγου και νομίζω ότι ήδη έχει αρχίσει αυτός ο οικονομικός διάλογος. Απόδειξη η σημερινή μας συνεδρίαση. Βέβαια, η πρόκληση είναι πώς αυτός ο οικονομικός διάλογος θα ενταχθεί σε μια κατάσταση που είναι δυναμική, που δεν είναι στατική και που αλλάζει ραγδαία. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά έχουμε και την πραγματικότητα που μεταβάλλεται συνεχώς, όπως έχουμε διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό. Και αυτή η πραγματικότητα βρίσκεται εκτός των θεσμικών οργάνων. Είναι πολύ δύσκολο να βρούμε το σωστό συνδυασμό, τη σωστή, το σωστό συμβιβασμό και να ταιριάξουμε στα χρονοδιαγράμματα αυτά τον οικονομικό διάλογο. Σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, αναφερθήκατε στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και διαπιστώστε μία ε, επιβράδυση αυτής της ανάπτυξης, όντως. Και απόφαση της ΕΚΤ για μείωση των επιτοκίων είναι απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να ε, διαχειριστεί αυτή την ε, ε, οικονομική κατάσταση που όλο και χειροτερεύει. Βέβαια, η μείωση των επιτοκίων δεν είναι η μοναδική λύση για την αποτροπή της επιδείνωσης. Βέβαια, και δεν θα είναι αποτελεσματική αν δεν εφαρμόσουν όλα τα κράτη-μέλη ε, φορολογικές πολιτικές λιτότητας. Πάντως, όπως είπε ο Επίτροπος Ρεν, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα υπέρογκου δημόσιου χρέους που το παρουσιάζουν ακόμη και χώρες που έχουν τριπλό αλφα στην αξιολόγηση πιστοληπτική τους εικονότητας και αυτό σε τελική ανάλυση δεν θα είναι βιώσιμο Πάντως, αυτή τη στιγμή θα είχε νόημα να υιοθετήσουμε πιο επεκτατικές πολιτικές σε χώρες που δεν αντιμετωπίζουν τόσο οξύ πρόβλημα δημοσιοχρέους. Πάντως, όπως είπε και ο Υπουργός Ροστόφης και πριν από λίγο, ελάχιστες σήμερα είναι οι χώρες στην Ευρώπη ε, που εφαρμόζουν κλασική και ισιανή πολιτική, όπου η Κεντρική Τράπεζα ε, δεν χρηματοδοτεί το δημόσιο χρέος. Και άλλωστε αυτή η δυνατότητα αποκλείεται από τι συνθήκες. Γι' αυτό και η κατάσταση είναι περίπλοκη. Και όλα αυτά τα διλήμματα θα ξανασυζητηθούν και σήμερα κατά πάσα πιθανότητα. αλλά και στην επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup. Και σήμερα μέχρι αργά το βράδυ και αύριο στο ΕΚΟΦΗΝ. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την σοβαρότητα της κατάστασης. Um, we've got now λοιπόν, έχουμε τώρα τους Σικλούνα ε, και Βέρνερ Λάγκεν. Θα σας ακούσουμε και τους δύο γιατί έχουμε μείνει μόνο πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Ούντο. Σε πολλές ε, περιπτώσεις και στην τελευταία αλλαγή της συνθήκης πάντα αναφερόμαστε στο ευρώ σύνολο. Όταν μιλάμε λοιπόν για την οικονομική πολιτική, γιατί δεν αναφερόμαστε στην Ευρωζώνη στο σύνολό της. Ακούσαμε μόλις τον Όλη Ρεν να λέει πως να ξεπερνάμε το 90% του το χρέο σε κάποιες χώρες οπωσδήποτε δεν είναι ο σωστό δρόμο κτλ. Συμφωνούμε όλοι, αλλά γιατί χώρες όπως η Ελλάδα και οποιαδήποτε άλλη χώρα που ξεπερνάει αυτό το ποσοστό να ε, θεωρηθούν ως το σημείο αναφοράς. Ο λόγος για τον οποίο η G20 το ΔΝΤ δυσκολεύεται να χρηματοδοτήσει την Ευρωζώνη λένε πως κοιτάνε την ε, Ευρωζώνη στο σύνολό της. Έχουν ε, ισοζύγιο συναλλαγών, θετικό, μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, χρέο χαμηλότερο από την Ιαπωνία. Οπότε, αν μιλάμε για ανάπτυξη, είτε μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, πρέπει να βλέπουμε την Ευρωζώνη συνολικά. Και όταν το αποφασίσουμε αυτό, μετά πρέπει να δούμε ποια χώρα μπορεί να πληρώσει το οτιδήποτε. Γιατί υπάρχουν χώρε που μπορούν να έχουν την πολυτέλεια κάποιων ε, σχεδίων απασχόλησης, άλλες δεν μπορούν. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέω. Δεν μπορούμε να παίρνουμε τις χώρες που ξεπερνάνε το 90% ή το 100% ως σημείο αναφοράς και να κρύβουμε πίσω από αυτές ε, τις υπόλοιπες και να λέμε δεν μπορούμε να πληρώσουμε το χ και το ψ. Βέρνερ. Ναι. Θα ήθελα να στηρίξω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπούλμαν το γεγονός πως ειδικά στην κρίση του ευρώ δεν εφευρέθηκαν μόνο νέα μέσα, αλλά θεωρούμε είτε γιατί δεν εμπιστευόμαστε την Κομισιόν, είτε θέλουμε να εμποδίσουμε το Κοινοβούλιο από το να μιλήσει, είτε γιατί χρησιμοποιούμε τη δικαιολογία πως η νομοθετική διαδικασία διαρκεί πάρα πολύ, έχει γίνει κανόνας η διακυβερνητική μέθοδος. Αυτό είναι λάθος η κοινοτική μέθοδος χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ και για δημοκρατικούς λόγους και αν δείτε το τι έχει γίνει σε όλες τις συνόδους τους τελευταίους 15 μήνες είχαμε μια κομισιόν ενεργή η οποία έκανε τις προτάσεις τηρώντας την ε, συνθήκη της ε, Λισαβόνας ακριβώς λόγω της δημοκρατικής νομιμοποίησης που προκύπτει από το έρετο κοινοβούλιο και την συναπόφασή του και με τη διπλή πλειοψηφία του Συμβουλίου και των κρατών και του πληθυσμού δηλαδή και λέει πως αυτή η διαδικασία πρέπει να ακολουθεί. Εν τω μεταξύ αυτή η διαδικασία έχει παραγωνιστεί τόσο ώστε θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως η Λισαβόνα πηγαίνει προς αποτυχία εάν οι Υπουργοί δεν τηρούν τις υφιστάμενες συνθήκες. Και το ότι η Κομισιόν το προσπερνά αυτό χαλαρά. Το ξέρουμε εδώ και το ξέρουμε σε πολλές περιπτώσεις. Παραδείγματο χάρη η Σουηδία που δεν έχει opt-out από την Ευρωζώνη, η Σουηδία δεν ε, προειδοποιείται από την Κομισιόν να παραμείνει εκτός μόνο η Δανία και η Μεγάλη Βρετανία έχουν κάνει το opt-out και αυτό για μένα είναι σκάνδαλο. Συν το ότι το άρθρο 122 πλέον έχει τεντωθεί, έχει φτάσει στα όρια του για να βρεθεί ένας τρόπος ο οποίος θα ήταν διακυβερτικός. Εάν είναι να παραμείνει μια κοινότητα δικαίου η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η κατάσταση δεν είναι πλέον ανεκτή. Και θα πρέπει να τα ακούσουν αυτό οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων και ο... η Προεδρία, η Πολωνική είναι σε δύσκολη κατάσταση όσο παραδείγματο χάρη στον ε, κανονισμό χρηματαγορών μόνο μπλοκάρει η Μεγάλη Βρετανία και δεν χρησιμοποιούμε τον κανόνα της ε, διπλής ε, πλειοψηφίας για να ξεπεράσουμε το ζήτημα. Δεν φταίει η Πολωνία, φταίνε οι υπόλοιπε χώρες μέλη. Uh, Ευχαριστώ πολύ για, αυτή ε, για αυτές τις ερωτήσεις. Επί του πρώτου ερωτήματος μπορώ να απαντήσω δεν ε, είναι ότι ε, τα θεσμικά όργανα δεν βλέπουν σαν σύνολο την ε, οικονομική αγορά, αλλά πρέπει να πιστούν ε, οι αγορές. Το δύσκολο είναι αυτό, το να πείσουμε τις ε, αγορές. Και πιστεύω ότι μετά την κρίση και μετά την μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, θα είμαστε πιο κοντά σε αυτό το ιδεώδες. μιας πραγματικά κοινή ε, ζώνης ευρώ. Και τότε το ερώτημα θα απαντηθεί θετικά, θα μπορεί να απαντηθεί θετικά. Για την ώρα, όπως είπα και προηγουμένως, είχαμε τοπιστατικές αγορές ε, βλέπουν την Ευρώπη και την Ευρωζώνη ε, σαν ναι μία ζώνη που έχει το ίδιο νόμισμα αλλά ε, που έχει διαφορετικούς οικονομικούς δείκτες, διαφορετικό χρέος και τα λοιπά. Και είναι δύσκολο να τους πείσουμε για το αντίθετο. Και ούτως ή άλλως και για την ίδια την Ευρώπη είναι δύσκολος ο χειρισμός μιας τέτοιας κατάστασης και είναι δύσκολο και για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ε, είναι ιδιαίτερως περιπεπλεγμένη η κατάσταση. και τα όσα συμβαίνουν σε μερικές χώρες ε, τώρα ε, είναι ένα σκέλος μονάχα της περιπλοκότητας ε, της κατάστασης. Εάν μετά από κάποια χρόνια, μετά από δέκα χρόνια... Area which, which is optimal. Ε, βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Θα πρέπει να βελτιωθούμε όσον αφορά το κοινό νόμισμα. Η δεύτερη ερώτηση ήταν μία άποψη ότι η κοινή προσέγγιση, κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ε, σε διάφορα ζητήματα είναι καλύτερη από την διακυβερνητική προσέγγιση. Βεβαίως ε, μπορώ να συμφωνήσω με μια τέτοια δήλωση. Όμως πιστεύω ότι απορρέει από την παρούσα δομή των συνθήκων και βεβαίω αντικατοπτρίζει και τη διαφορά ανάμεσα στην Ευρωζώνη και τις χώρες που δεν ανήκουν σε αυτήν. Σχετικά με το opt-out όσον αφορά το, το ευρώ, ε, κοιτάξτε, ξέρουμε πώς έχει η κατάσταση Είμαστε υποχρεωμένοι να μπούμε στην Ευρωζώνη. Είμαστε ήδη νομικά ε, ε, στην Ευρωζώνη, αλλά ε, με κάποια εξαίρεση. Και χωρίς το opt-out δεν έχει καμία έννοια το όποιο δημοψήφισμα γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε συμφωνήσει να μπούμε στην Ευρωζώνη το 2004, όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχαμε το καθεστώς της χώρας ε, που θα εγκρίνει κάποια στιγμή το ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Οδηγούμαστε λοιπόν στην ολοκλήρωση ε, της ακρόασης. Ούτως ή άλλως να υπενθυμίσω ότι το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ευρώ και ότι ακόμα και οι χώρες οι οποίες δεν είναι ακόμα μέλη έχουν το δικαίωμα ε, να μπουν στο ευρώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που καθίσατε και απαντήσατε στις ερωτήσεις. Και περνάμε τώρα στο υπόλοιπο, ε, στα υπόλοιπα σημεία της ημερήσιας διάταξής μας. Προχωράμε λοιπόν στο σημείο 4. Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα θέμα για το οποίο είμαι εισηγήτρια. Μια και δεν ε, έτσι, προκάλεσε τρομερό ενθουσιασμό το θέμα αυτό, το ανέλαβα εγώ θα ήθελα να κάνω μια πάρα πολύ σύντομη εισαγωγή. Γνωρίζω ότι υπάρχει εκπρόσωπος της Eurostat που εδώ που μπορεί να μας ε, πει δύο λόγια παραπάνω. Θα ήθελα να πω δύο λόγια λοιπόν και μετά να δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους της Eurostat και στους σκιώδεις εισηγητές. Η πρόταση αυτή αφορά αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εθνικών και Περιφερειακών Οργανισμών του 1995. Το κείμενο αυτό βασίζεται στην ε, τελευταία αναθεώρηση ε, των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά το σύστημα ε, των εθνικών λογαριασμών του 2008. Απλώς προχωράει σε περισσότερη λεπτομέρεια από ότι το αντίστοιχο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Το κείμενο απαρτίζεται από τον ίδιο τον κανονισμό και δύο παραρτήματα. Στο παράρτημα 1 υπάρχει η μεθοδολογία, ταξινόμηση και ε, οι κανόνες ε, όσον αφορά τους λογαριασμούς και στο παράρτημα 2 αναφέρεται η μεθοδολογία μεταβίβασης ε, των πληροφοριών. Ε, στο, το παράρτημα Α δεν μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα, ενώ η εργασία για το παράρτημα 2 ε, ακόμα συνεχίζεται και δεν θα ολοκληρωθεί πριν μερικού μήνες. Ε, είναι ε, πολύ τεχνικό το κείμενο και αρκετά μεγάλο, αρκετά μακροσκελές, ε, αλλά βεβαίως έχει και μεγάλη πολιτική σημασία. Αυτό που προτείνω να κάνουμε είναι να θεωρήσουμε, να το θεωρήσουμε σαν ένα πλαίσιο και να το δούμε θετικά περιμένοντας βεβαίως να έχουμε και περισσότερες πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή. Να δούμε δε ε, ε, κυρίως ε, τι κάνει το, τι κάνει το Συμβούλιο όσον αφορά τους διάφορους πίνακες. Να πω επίσης τα ε, στο παρελθόν, οι δαπάνες, ε, οι στρατιωτικές ε, και για την έρευνα και την ανάπτυξη το, δεν συνυπολογίζοντας το ΑΕΠ. Έχουμε λοιπόν μια αύξηση της τάξης του 2%. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ως αποτέλεσμα αυτής της συμπερίληψης. Όσον αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξης, ε, μου ζητήθηκε ε, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εάν είναι δυνατόν ε, να υπάρξει πρώτερη διαβούλευση έτσι ώστε κατά την άποψή τους όλες οι κατεξακολούθηση πράξεις κατεξουσιοδότης συγγνώμη πράξης να έχουν και οικονομική λογική αλλά βεβαίως θα πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν να δώσουμε ε, ρόλο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί θεσμικά δεν μπορούν ε, να ε, συνδιαβουλευθούν. Θα πρέπει να δούμε θεσμικά πώς μπορεί να γίνει. Επίσης, στο παράρτημα Β, στην μεταβίβαση των δεδομένων. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο μας ενδιαφέρει, ποιος θα έχει τα στοιχεία, πώς και πότε γίνεται λόγος, γίνεται ε, αναφορά σε 85 μέρες, ε, ενώ ε, εμείς τις η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει μείωση του χρόνου αυτού, 80 μέρες ενδεχομένως, γιατί θέλουν να έχουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τις πληροφορίες. Όμως αυτό το θεωρεί μεγάλο άχθος, το θεωρούν μεγάλο άχθος τα κράτη. Προσωπικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τα στοιχεία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Τέλος, έχουμε την επιλογή για τα ε, στοιχεία τα οποία θα συλλέγονται. Ε, υπήρχε μια, ε, ένα κείμενο ε, της ε, Στατιστικής Υπηρεσίας ε, του 93 σχετικά με την συλλογή στοιχείων του 95. γίνεται, εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε ποια είναι τα στοιχεία, πώς θα συλλέγονται και ποια είναι η δυνατότητα αντίθεσης που έχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτά είναι τα κυριότερα στοιχεία της έκθεσης. Βλέπω ότι έχουμε και τους σκιώδεις ηγητές εδώ. Θα δώσουμε αμέσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, εάν βεβαίως επιθυμούν να πάρει, επιθυμεί να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ λακωνικός γιατί καλύψατε πολλά σημεία. Όπως είπατε, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών προβλέπει το μεθοδολογικό πλαίσιο για την δημιουργία εθνικών λογαριασμών στην Ευρώπη. Και οι εθνικοί λογαριασμοί χρησιμοποιούνται για πολύ σημαντικέ ευρωπαϊκέ πολιτικέ, όπω είναι η πολιτική των ιδιών πόρων, η κατανομή των διαρθρωτικών κονδυλίων, το σύμφωνο σταθερότητα και ε, ε, ε, Σταθερότητα και ανάπτυξη, καθώ και για την δημιουργία κάποιων οικονομικών αναλύσεων. Η αναθεώρηση αυτή δεν προποθέτει και 15 χρόνια μετά την έγκριση του πρώτου κανονισμού για την ΕΣΑ, δεν προϋποθέτει κάποιες αλλαγές στην ε, θεμελιώδη δομή των λογαριασμών και η μελέτη επιπτώσεων, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, που πραγματοποιούσαμε, καταλήγει σε έναν υπολογισμό αύξησης 2% στο επίπεδο του ΑΕΠ μετά τις αλλαγές ε, που θεσπίσαμε. Οι βασικές αλλαγές που προτείνουμε, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι η κεφαλαιοποίηση του, της έρευνας και ανάπτυξης, η κεφαλαιοποίηση των στρατιωτικών δαπανών, η τα αγαθά προς, ε, τα εμπορεύσιμα ε, χρησιμοποιούνται με τη βάση της ε, ιδιοκτησίας και πιο λεπτομεριακή ανάλυση των συνταξιοδοτικών συστημάτων μέσω ενός συμπληρωματικού πίνακα που βελτιώνει τη συγκρισιμότητα των στοιχείων αυτών. Σε τεχνικό επίπεδο υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τις μεθοδολογικές αλλαγές, το επισημάνατε κι εσείς, ενώ κρεμεί η συζήτηση για το πρόγραμμα μεταβίβασης των δεδομένων. Βέβαια, έχουμε κάποια κατανόηση για τη θέση των κρατών μελών που σε πλαίσιο οικονομικής χρηματοπιστωτικής κρίσης και περικοπών στον προϋπολογισμό προτιμούν να είναι πιο επιφυλακτικά σε ό,τι αφορά τι απαιτήσει μα για το πρόγραμμα μεταβίβαση δεδομένων. Πάντω, η Eurostat πιστεύει ότι μια καλύτερη παρακολούθηση των ε, νομισματικών αλλαγών και των οικονομικών αλλαγών τα επόμενα 15-20 χρόνια προποθέτει ρεαλιστικά προγράμματα αλλά και φιλόδοξα προγράμματα μεταβίβαση δεδομένων και προσβλέπουμε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μείνουμε στο φιλόδοξό μα πρόγραμμα. Θέλουμε να περιορίσουμε τον αριθμό των εξαιρέσεων και παρεκκλήσεων που ζητούνται από τι χώρε μέλη και ευελπιστούμε ότι θα συμπεριληφθούν κάποια στοιχεία όπως είναι η κεφαλαιο κεφαλαιοποίηση ε, τη έρευνα και ανάπτυξη, καθώ και οι πληροφορίε για τι συντάξει θα τύχουν τις υποστήριξή σα. Είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για να βελτιώσουμε τα δεδομένα που έχουμε για την οικονομία μας. και όπως φάνηκε και τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν αρκετά κενά και πολλές αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνουμε πληροφορίες για την οικονομική μας ανάπτυξη. Και ελπίζουμε την τελευταία πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεωρημένη ΕΣΑ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικό και Περιφερειακό Λογαριασμό 2010, θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Θα ήθελα επίσης ε, να προσθέσω ένα από τα στοιχεία που επισημάνατε, τη κατεξουσιοδότηση πράξη. Προτείναμε εκτεταμένη χρήση κατεξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό λόγω τη ταχύτητα και τη ραγδαία εξέλιξη των οικονομικών αλλαγών. Γι' αυτό και εμεί χρειαζόμαστε έναν ταχύ τρόπο ενημέρωση των μεθοδολογικών απαιτήσεων για την ε, παραγωγή των δεδομένων εθνικών λογαριασμών. Τα κράτη-μέλη δεν είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδη για την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι η Eurostat προτείνει έναν ελαστικό τρόπο για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας και του τρόπου μεταβίβασης δεδομένων. Εξού και η πρότασή μας και προσβλέπουμε και στην δική σας υποστήριξη. Φυσικά έχουμε πολλούς και διάφορους τρόπους για την ε, συμπερίληψη και το διάλογο με την ΕΚΤ. Έχουμε καθημερινή ε, επαφή με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για όλα τα στατιστικά μας δεδομένα, οπότε θα επιληθεί και αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε εκπρόσωπο και του Συμβουλίου που ζήτησε το λόγο. Συνήθως ε, δεν ε, το κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά αν μου υποσχεθείτε δεν θα με ακρηγορήσετε δεν έχω αντίρρηση να κάνω μια μικρή εξαίρεση. Ποιος θα λάβει το λόγο εκ μέρους του Συμβουλίου. Κανείς. Dziękuję bardzo Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την κατάσταση των πραγμάτων και σε τι φάση βρισκόμαστε στο Συμβούλιο. Και μπορώ και να σας στείλω και γραπτώ σε αυτή τη, αυτές τις πληροφορίες. Κάποιες ε, πληροφορίες πάντως για τα θέματα που θίξατε σήμερα. Σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες ε, μεταβίβασης δεδομένων, όπως ε, προσδιορίστηκε στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, οι συζητήσεις αυτές θα γίνουν αργότερα, αναβλήθηκαν, δεν έχουν ε, ληφθεί αποφάσεις σχετικά για τις προθεσμίες, γιατί πρόκειται για οριζόντια θέματα και θα συνδυαστούν με, την, με τις αποφάσεις για τους πίνακες. Σε ό,τι αφορά το παράρτημα Β, συνεχίζουμε τις συζητήσεις για τους πίνακες. Σε ό,τι αφορά τις παρεκκλήσεις τώρα, τις εξαιρέσεις που ζητούν οι χώρες μέλη, και η συζήτηση αυτή αναβλήθηκε για μεταγενέστερη συζήτηση μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος ε, μεταβίβαση δεδομένων γιατί τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν έτσι να επαληθεύσουν τα προκαταρκτικά του συμπεράσματα και τις αιτήσει για τις παρεκκλήσεις και να συνεχίσουν τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά για το ουσιαστικό τμήμα της συζήτησης, ε, δεν προλάβαμε ακόμη να εγγύψουμε στα ουσιαστικά ζητήματα. Γι' αυτό δεν έχουν μπηθεί σχετικέ αποφάσεις. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεοδόρ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω πως είναι μια καλή στιγμή να αναβαθμιστεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών και αν θεωρούμε πως με τον νέο μας κανονισμό όσον αφορά την οικονομική αυτή διακυβέρνηση υπάρχει κάποιο συσχετισμός μεταξύ αύξησης του ΑΕΠ και αύξηση των δημοσίων δαπανών τότε μπορούμε να δούμε πως έχουμε σημειώσει προόδο και βασιζόμαστε πάρα πολύ στην οικονομική μας πολιτική, στην ακαιρεότητα και την ορθότητα των δεδομένων των εθνικών λογαριασμών. Οπότε νομίζω πως είναι καλή στιγμή για να αναβαθμίσουμε τη μεθοδολογία αυτή. Νομίζω πως είναι θετικό επίτευγμα το ότι διατηρήσαμε την αρχή το να χρησιμοποιούμε αυτούς τους δορυφορικούς λογαριασμούς για να καταγράφουμε όλα τα είδη δραστηριοτήτων που δεν μπορούν να εκφραστούν με χρηματικούς όρους και έγιναν πολλές συζητήσεις π.χ. για τη ρήπανση, το πώς μετράμε την ευημερία στο κάθε κράτος μέλος. Νομίζω πως ακόμα και αν το Συμβούλιο είχε ήδη συμφωνήσει σε αυτό το παράρτημα Α, νομίζουμε πως στις συζητήσεις μας αυτές για το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Στατιστική Επιτροπή θα έπρεπε να ψάξουν περαιτέρω ειδικά τον πληθωρισμό το πώς λαμβάνεται υπόψη είναι ο πληθωρισμός στο ΑΕΠ γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ πληθωρισμού κατανάλωσης ε, των πολιτών και αυτό το οποίο λέμε ε, από πληθωρισμός του ΑΕΠ. Και όταν έχουμε ανάπτυξη 1-2% και πληθωρισμό της τάξης του 2-3% τότε οποιοδήποτε σφάλμα στον υπολογισμό του πληθωρισμού ε, έχει σημαντικό αντίκτυπο στο επίπεδο του ΑΕΠ. Νομίζω επίσης πως θα πρέπει να ερευνήσουμε περαιτέρω το πώς αντικατοπτρίζεται στους εθνικούς λογαριασμούς, πώς αντικατοπτρίζονται οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και επίσης νομίζω πως δεν χρησιμοποιήσαμε αρκετά τα αποτελέσματα του κοινωνικού λογιστικού συστήματος για να αναλύσουμε το τι συμβαίνει στην εξέλιξη των τομεακών αυτών λογαριασμών. Ωραία, αναμένουμε την έκθεσή σας και θα συνεργαστούμε βεβαίως. Σας ευχαριστώ Έντουαρτ. Ευχαριστώ πολύ Σάρον. Οπωσδήποτε μια αναθεώρηση θεμελιωδών στατιστικών στοιχείων όπως η ε, εθνική και περιφερειακή λογαριασμή μετά από 15 χρόνια είναι βεβαίως κάτι το ευπρόσδεκτο. Έχει γίνει πολλή δουλειά στον ΟΗΕ αλλά υπάρχει βεβαίως μια κάποια σχέση ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να προσαρμόσουμε ε, τις αναθεωρήσεις αυτές, τις ανάγκες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς βεβαίως να αντιβαίνουμε κάπου το σύστημα του ΟΗΕ. Από πλευρά χάραξης πολιτικής, το ΑΕΠ, όπως επισημάνατε, είναι ένα μέτρο σύγκριση που χρησιμοποιείται, είτε μιλάμε για τα δημόσια οικονομικά, ανάπτυξη, πληθωρισμό κτλ. Οπότε είναι κρίμα το ότι χωρίς να το ότι δεν συνειδητοποιούν πολύ ότι είναι ε, ένα τελές μέτρο σύγκρισης που δεν συμπεριλαμβάνει κάποιες δραστηριότητες όπως τις δραστηριότητες στα νοικοκυριά μετρά τον δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος τομέας σε πολλές χώρες βεβαίω είναι πολύ εκτεταμένος μεταξύ 30 και μέχρι και πάνω από 50% του ΑΕΠ αλλά δεν μετράει καθόλου τις εκροές, μόνο τις εισρωές. Δηλαδή η λιγότερο αποτελεσματική ε, δημόσιοι τομείς που απασχολούν περισσότερους και παράγουν λιγότερα ε, φαίνονται ως να αποτελούν ένα τομέα ανάπτυξης. Ενώ δεν είναι. Ενώ αυτοί που είναι πιο αποτελεσματικοί και ε, απασχολούν λιγότερους δεν φαίνεται πουθενά οι επιδόσεις τους στους εθνικούς λογαριασμούς. Το ίδιο και για το περιβάλλον δεν βλέπουμε στους εθνικούς λογαριασμούς ε, μια πτυχή περιβαλλοντική. Μιλάμε για πράσινες δουλειές, ε, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε τον παραδοσιακό τομέα των κατασκευών και παρά το ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πιλωτικά έργα από την Eurostat και τον ΟΣΑ, ελπίζω να συμπεριληφθούν ε, στον τομέα των κατασκευών και της βιομηχανίας. Μια υποκατηγορία για τις πράσινες θέσεις εργασίας θα βοηθήσει ειδικά την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει τους τομείς εκείνους που είναι υποσχόμενοι για το μέλλον. Οπότε, γενικά, καλώς ορίζουμε τις αναθεωρήσεις αυτές, αλλά αναμένουμε την έκθεση αυτή, γιατί και εγώ ως σκιώδης βεβαίως είμαι έτοιμος να βοηθήσω και εσάς κυρία Πρόεδρε και τους υπολείπους για να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση. Σας ευχαριστώ. Όπως είπα, τον έλαβα ως πρόεδρος, ελπίζοντας βέβαια θα με βοηθήσουν και οι αντιπρόεδροι. Στόχος μας είναι να καταρτήσουμε την, το σχέδιο έκθεσης ήδη το Δεκέμβριο με προθεσμία για τις τροπολογίες την 18 Ιανουαρίου, ώστε να το συζητήσουμε τέλη Φεβρουαρίου και να ψηφίσουμε 20 Μαρτίου και στην πρώτη ορομέλεια του Μαΐου. Αυτές είναι, αυτή είναι η στόχη μας με τους αντιπροέδρους και θέλουμε να συμπεριλάβουμε ήδη στο, στην έκθεση όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα και να έχουμε και κάποιο χρόνο να χτενίσουμε και τα υπόλοιπα θέματα ανάλογα με τις συζητήσεις. Πέραμε στο επόμενο σημείο, το 5, φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και του ηλεκτρισμού. Η συγγήτριά μα για το σημείο αυτό είναι η Astrid, Λούλινγκ. Ο Φίλιπ Λάμπερτ ε, ζήτησε συγγνώμη γιατί κόλλησε κάπου αλλού, δεν μπόρεσε να είναι στην προηγούμενη συζήτηση, ούτε τώρα. Αστρίτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στις 31 Αυγούστου συγγνώμη, είχα εξηγήσει ότι με την αναθεώρηση της οδηγίας για την φορολογία των ενεργειακών προϊόντων τον Απρίλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κάτι πολύ πιο περίπλοκο από ένα απλό καλοπισμό ενός προϋπάρχοντος κειμένου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε με την αναθεώρησή της μια πραγματική επανάσταση Κοπέρνικου με άμεσες αλλά και βραχυπρόθεσμες συνέπειες. Εγώ ασχολήθηκα με την πρόταση αυτή επισημένοντας κάποιες αντιφάσεις της αναθεώρησης και φυσικά είπα ότι περιμένω την ε, βοήθεια των συναδέλφων, είτε είναι σκιώδηση ή όχι. Και μετά από εντατική ενασχόληση με το θέμα αυτό και επαφές με εκπροσώπους ε, των Υπουργείων, των Τελωνίων, εκπροσώπων επαγγελματικών κλάδων της κοινωνίας των πολιτών. Ε, όλοι πιστήκαμε από τη σημασία του κειμένου, αλλά Δυστυχώ ο τρόπος που ερμηνεύουν το κείμενο οι διάφοροι φορείς είναι διαφορετική. Γι' αυτό και μετά από διαπίστωση όλων αυτών των αντιφάσεων αποφάσισα να περιμένω λίγο πριν υποβάλω ένα ισορροπημένο και συνεκτικό κείμενο που να χρησιμοποιηθεί και ως βάση συμβαστική λύση από το Συμβούλιο. Τώρα με το σχέδιο γνωμοδότησης, με το σχέδιο έκθεσής μου πιστεύω ότι έχουμε μία ε, με στη βάση και ευελπιστώ ότι θα τύχει τη υποστήριξη των συναδέλφων που φαντάζομαι όμως θα υποβάλουν και τροπολογίες και άλλες τροπολογίες. Επί της αρχής, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η παρούσα πρόταση αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής 2020-2020 σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και από την άποψη αυτή πρόκειται για ένα κεφαλαιόδες, ε, θεμελιώδες κείμενο. Αλλά ας μην ξεχνούμε ότι η φορολογία των ενεργειακών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε, ε, σε, κλιματικά, σε κλιματικές ή περιβαλλοντικές απαιτήσεις, παρόλο που αυτές είναι πολύ σημαντικές. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής καθώς και οι στόχοι της ε, βιομηχανικής πολιτικής ε, αποτελούν πολύ σημαντικά διακυβεύματα. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αναζητήσουμε και να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αντιφατικών μερικές φορές ε, στόχων, προκειμένου να δώσουμε τη σωστή όθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό επιχείρησα και εγώ με την έκθεσή μου και με τις προτάσεις που κατέθεσε εκεί. Ακολουθώντας τον ίδιο ρυθμό, θα ήθελα να πω ότι κρίνω σκόπιμο να φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη συνάφεια και συνέπεια μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που άπτονται τις ενέργειες και που αποτελούν αντικείμενο εξέταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο. Για παράδειγμα, έχουμε την οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα αυτή τη στιγμή εξετάζεται από άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν να συντονιστούμε και να συμφωνήσουμε σε ό,τι αφορά τους ε, θεμελιώδεις προσανατολισμούς μιας πανευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής που ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί. Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται σε ευσεβείς πόθη, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα ε, να τους ε, επισημάνουμε. Τώρα επανέρχομαι στο κείμενο. Εγώ προτείνω να στηρίξουμε τη μεθοδολογική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να φορολογήσει με διπλή βάση την ενέργεια, με βάση την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα και με βάση το ενεργειακό περιεχόμενο του προϊόντος. Το διπλό αυτό σύστημα φαίνεται και πιο λογικό, αλλά και πιο συνεπές και συνεκτικό από το προηγούμενο. Γιατί διευκολύνει την καλύτερη χρήση των ενεργειακών πόρων και ενισχύει την ε, αυξημένη χρήση των ε, λιγότερο ε, ρηπογόνων ενεργειακών πηγών. Είμαι υπέρ αυτής της προσέγγισης. Άλλωστε, η, η εισαγωγή του φόρου, 20, φόρου διοξιδίου του άνθρακα 20 ευρώ τον τόνο ε, ανατόνο διοξιδίου του άνθρακα θα εξασφαλίσει φορολογικά έσοδα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020. Διόλου αμεληταίο ποσό σε τόσο χαλεπούς δημοσιονομικούς καιρούς που διανύουμε. Πάντως, ένα από τα πιο απτά στοιχεία της νέας πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή ε, η ανάγκη σεβασμού από τα κράτη-μέλη της ε, αναλογικότητας μεταξύ των διαφόρων ελάχιστων ορίων που θεσπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν με βρίσκει σύμφωνη. Είχα εκτενέστατες διαβουλεύσεις για το θέμα αυτό. Βέβαια σημείωσε τη θέση και των κρατών μελών. Με εξαίρεση 3-4, όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ε, εξέφασαν την αντίθεσή τους με το θέμα αυτό. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πολιτική πραγματικότητα. Και ακόμη και αν ε, δεν ισχύει εδώ διαδικασία συναπόφασης, θεωρώ ότι ο ρόλος μας δεν είναι να προτείνουμε κάτι που δεν έχει καμία πιθανότητα να εγκριθεί, μια και προσκρούει διαφωνία της πλειοψηφίας των κρατών μελών. στόχος μας είναι και νομίζω ότι καθήκον μας είναι να προτείνουμε συμβαστικές προτάσεις που θα γίνουν αποδεκτές από το Συμβούλιο. Ακόμη κι αν έτσι ρίξουμε λίγο νερό στο κρασί μας και αμβλύνουμε κάπως τις αρχικές φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τώρα το θεσμικό επίπεδο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο αυστηρός ε, σεβασμός και η αυστηρή τήρηση της αναλογικότητας ε, από τα κράτη-μέλη θα έχει επίδραση στο επίπεδο φορολογίας ε, των διαφόρων ενεργειακών προϊόντων στις 27 χώρες μέλη. Ενώ μέχρι στιγμής ίσχυε η αρχή των ελάχιστων κατοφλίων Πάντως, η αρχή της αναλογικότητας στην πράξη θα έχει σημαντικές αποσταθεροποιητικές συνέπειες. Και η πιο περίτρανη απόδειξη θα είναι η σημαντική αύξηση της τιμής του ντίζελ στην συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μέλων. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα ακρεφνούς εφαρμογής αρχής της αναλογικότητας. Τώρα, από πολιτική άποψη η σημαντική αύξηση της τιμής του ντίζελ στις περισσότερες χώρες μέλη. Για να σας δώσω ένα μόνο παράδειγμα, στη Γερμανία η αύξηση θα είναι της τάξης του 31 cents ανά λίτρο ε, μέχρι το 2023. Ε, μια τέτοια αύξηση θα δημιουργήσει και το μέτρο αυτό θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιλύει. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο μπροστά σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τις άλλες περιοχές του κόσμου που σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την τεχνολογική ανάπτυξη των κινητήρων δίζελ. Και η τεχνολογική αυτή ανάπτυξη προϋποθέτει ε, έρευνα εχμής και αυτή η προηγμένη έρευνα, τεχνολογική έρευνα ε, συνιστά το βασικό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις υπόλοιπους οικονομικούς εταίρους. Με βάση όλα αυτά τα κριτήρια δεν νομίζω ότι είναι λογικό να επιβάλλουμε στην ευρωπαϊκή μας αυτοκίνητο βιομηχανία που ήδη αντιμετωπίζει έναν λησαλέοντα ανταγωνισμό από τρίτες χώρες και αντιμετωπίζει και διαρθρωτικά προβλήματα, δεν κρίνω να τις επιβάλλουμε και τον κλονισμό αυτό και το πλήγμα αυτό που θα την αποσταθεροποιήσει. Ακόμη και η δεκαετής μεταβατική περίοδος δεν αρκεί για να ε, μειώσει τα αρνητικά αποτελέσματα. Τρίτο ουσιαστικό επιχείρημα που αντιτάσσεται στην εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας αφορά την επίπτωση που θα έχει στις τιμές κατανάλωσης. Ε, ο πληθωριστικός κίνδυνος ε, εξαιτίας αυτής της σημαντικής αύξησης της τιμής πολλών καυσίμων δεν είναι εύκολο να αποσοβηθεί και πολλές χώρες μέλη Εξαιτία ακριβώ τη δεινή οικονομικής κατάστασής τους και πριν από λίγο το σχολιάσαμε, δεν θα μπορέσουν να μειώσουν τους φόρους ε, που επιβάλλονται στην κατανάλωση βενζίνης. Οι καταναλωτές λοιπόν θα δεχτούν και αυτοί ένα πλήγμα από την αρχή της ε, αναλογικότητας, όπως ε, και ο, ο, ο τομέας των μεταφορών και ιδιαίτερα οι δημόσιες συγκοινωνίες που ε, θα δουν το κόστος λειτουργίας να αυξάνεται. γιατί η εξελίξη των ημών ενεργειακών προϊόντων αποτελεί μια, αποτελεί μια σημαντική αιστεία πληθωρισμού. Μεταξύ του 13 και του 16% είναι υπολογισμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί έχουμε ε, αύξηση του πληθωρισμού πάνω από 30% εξαιτίας ακριβώς της αύξησης των τιμών ε, του πετρελαίου. Μέσα σε ένα χρόνο οι τιμές ε, πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 13 με 16%. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους θα πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε την εφαρμογή μηχανισμών που θα τροφοδοτήσουν αύξηση των τιμών και άρα πληθωρισμό. Ως εκ τούτου λοιπόν προτείνω να διαγράψουμε αυτή τη διάταξη που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εφαρμογή, ακρεφνή εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας. Επίσης αντιτάσσομαι κάθετα στην πρόταση αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των ελάχιστων κατοφλίων ε, φορολόγησης στις ε, εξελίξεις των τιμών ε, ή στην βασική τιμή του διοξιδίου του άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Πρόεδρε, που σπέβδει να καταδικάσει την αυτόματη, τη αριθμική αναπροσαρμογή των μισθών, όπου υπάρχει ακόμη, με τα ίδια επιχειρήματα, ελαφρά την καρδία, εισάγει αυτή την αυτόματη, τη αριθμική αναπροσαρμογή στη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό ο νομοθέτης να έχει τον τελευταίο λόγο για τα θέματα αυτά και μία ε, τιμαριθμική αναπροσαρμογή δεν είναι σκόπιμη εδώ. Περιμένω φυσικά και τη γνώμη των υπόλοιπων σκιωδών εισηγητών αλλά και των λοιπόν συνοδέλφων αλλά προηγουμένως να σταθώ σε ένα σημείο που αφορά τα καυσίματα, τα καύσιμα υποκατάστασης ε, ε, και νομίζω ότι για λόγους συνέπειας τα ίδια επίπεδα φορολογία, οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστέ που στηρίζονται στο ενεργειακό περιεχόμενο και στο, στην επίπτωση διοξιδίου του άνθρακα να εφαρμόζονται για όλα τα καύσιμα, ακόμη και για το αέριο ε, υγροποιημένο πετρελαίου. Γιατί τα σχετικά πλεονεκτήματα κάθε καυσίμου σε ό,τι αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ε, ε, λαμβάνονται αυτόματα υπόψη από το φορολογικό καθεστώ. Κανένα άλλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν χορηγείται στην περίπτωση αυτή. Παρ' όλα αυτά και μια και το επίπεδο ε, ο ισχύων φορολογικό συντελεστής ε, στα αέρια αυτά είναι πολύ χαμηλό ή μερικέ φορέ ανύπαρκτο σε ορισμένα κράτη-μέλη. Θα χρειαστεί φυσικά κάποιο χρόνο πριν ε, εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα αυτών των αερίων ε, με τα συμβατικά καύσιμα εξαιτία των τεράστιων εξόδων που χρειάζονται σε επενδύσεις και υποδομές. Γι' αυτό θα έλεγα να περιορίσουμε την αύξηση του ελάχιστου κατοφυλίου σε αυτό που προβλέπεται από το 2015 και να, να μην την εφαρμόσουμε αυτή την προβλεπόμενη αύξηση από το 2018. Ένα τέτοιο περιορισμό τη αύξηση θα επιτρέψει αυτά τα υποκατάστατα καύσιμα να τύχουν ενός συγκριτικού πλέον εκτήματος ε, που είναι απαραίτητο για να ε, χρησιμοποιήσουν πιο ε, αποδοτικές οικονομικά τεχνολογίες για την ενέργεια. Επίσης, ήθελα να τονίσω ότι προσπάθησα να θετήσω μια ρεαλιστική προσέγγιση, γιατί ο φόρος διοξιδίου του άνθρακα για όλους τους τομείς που δεν, που δεν υπόκεινται στο σύστημα ε, εκπομπής, ε, εμπορίας ε, εκπομπών. Είναι πολύ σημαντικό και το να έχουμε μια μεθοδολογία για, την, για τον υπολογισμό των ελάχιστων κατοφλίων που εφαρμόζονται στις διάφορα, στα διάφορα ενεργειακά προϊόντα είναι σημαντικό. Παρόλο που πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη φορολογία με βάση τον όγκο, αντίθετα με την πρώτη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Είναι πολύ σημαντικέ όλε αυτέ οι αλλαγέ και προτείνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τις εγκρίνει και να τις υποβάλει στο Συμβούλιο. Δεν θα πρέπει να είμαστε ακραίοι ούτε προς την ούτε προς την άλλη κατεύθυνση γιατί διάβασα κάποιες γνωμοδοτήσεις, σχέδια γνωμοδότησης και πραγματικά έμεινα άναβη από τις ακρότητες που περιλαμβάνουν μπορεί ε, να γίνει κάπως πιο φιλόδοξη η δική μου έκθεση, θα εξαρτηθεί και από τις τροπολογίες, αλλά όχι τόσο ρίζοσπαστική όπως προτείνουν μερικοί συντάκτες γνωμοδότησης. Γιατί άμα υιοθετήσουμε τέτοιες ακραίες θέσεις, αποκλείεται η πρότασή μας να γίνει δεκτή από το Συμβούλιο. Πιστεύω ότι η πορεία των συζητήσεων και η έγκριση αυτής της έκθεσης θα μας επιφυλάξει πολλές εκπλήξεις. Πάντως, ελπίζω κάποια στιγμή να εγκριθεί αυτή η έκθεση. Και αυτή τη στιγμή δεν ασχολήθηκα με την εξαίρεση της ναυτιλίας ή της αεροπορίας Δεν περιλαμβάνω τίποτα για τις εξαιρέσεις αυτές στη δική μου έκθεση. Και απέφυγα και άλλα προβλήματα. Που όμως κάποια στιγμή αργότερα θα πρέπει να συζητηθούν. Όπως η εξαίρεση της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας, ηχθειοκαλλιέργειας, της δασοκο... της δασοκομείας, τα καύσιμα των οικοκυριών. Είναι πολλές και διάφορες οι εξαιρέσεις που προτείνονται και παραλαμβάνω δεν ασχολήθηκα με τα σημεία αυτά προς το παρόν. Και να σας ε, ενημερώσω και για κάτι που έμαθα σήμερα το απόγευμα. Το απόγευμα λοιπόν και λαμβάνοντας υπόψη τις αντιθέσεις ε, στο Συμβούλιο των Υπουργών, είναι πιθανό η Πολωνική Προεδρία να μην θίξει το ζήτημα, γιατί φαίνεται να είναι αδύνατη οποιαδήποτε επίτευξη συμβιβασμού. Και διαβάζω στο Financial Times της Γερμανίας πως ε, τα σχέδια της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, από ό,τι φαίνεται δεν θα εγκριθούν λόγω της αντίστασης των κρατών μελών. Στην συνεδρίαση των πρέσβεων πάρα πολλά κρατημέλη εξέφρασαν πάρα πολύ μεγάλες επιφυλάξεις για την ε, φορολογία των καυσίμων. Είναι αδύνατο να επιτευχθεί συμβιβασμός για τα σχέδια του Επιτρόπου κυρίου Σεμέτα για εναρμόνιση της ε, φορολόγησης της ε, ενέργειας. Υπάρχει μόνο περιορισμένη υποστήριξη από ό,τι φαίνεται είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές ώστε η συζήτηση που είχε προγραμματιστεί για ε, αύριο εννοεί σήμερα βεβαίως για ενημέρωση των Υπουργών Οικονομικών ε, κινδυνεύει να μην διεξαχθεί. Εγώ θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν αν αυτό ισχύει. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα αποτύχει η πρόταση σε μέτα στο Συμβούλιο και αν αυτό συμβεί θα πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε και τι προτιθέμεθα να κάνουμε με την έκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Άστριντ. Θα το παρακολουθήσουμε το ζήτημα. Ε, είναι εδώ πέρα οι περισσότεροι σκιώδεις ε, εισηγητές. Θα ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον ε, συνάδελφο, τον κύριο Σικλώνα. Ο κύριος Λούτβιχ, βεβαίως απουσιάζει, ζητεί συγγνώμη μου, έστειλε κάποιες σημειώσεις που θα διαβάσω. Συμφωνεί με κάποια στοιχεία του σχεδίου εκθέσεως και θεωρεί πως κάπου αλλού έχει αδυναμίες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τα θετικά. Θεωρεί πάρα πολύ καλό το ότι το βασικότερο στοιχείο της πρώτης κομισιόν γίνεται δεκτό, αυτή ε, φορολογική δομή που φασίζεται και στον στην περιεκτικότητα σε ενέργεια και στο διοξίδιο του άνθρακα. Και βεβαίως αυτό ε, είναι λογικό στο πλαίσιο μείωση εκπομπών και αύξησης εσόδων. Και βεβαίως η όθηση για να λειτουργήσει αυτή η οδηγία είναι κάτι το πάρα πολύ λογικό. Η ενέργεια είναι ένας τομέας όπου ε, εδώ και χρόνια έχουμε εξελίξεις, αλλά ο συντονισμός μεταξύ των ε, διαφόρων πρωτοβουλειών δεν ήταν αρκετά μεγάλος. Χρειάζεται μια πιο συνεκτική προσέγγιση και βεβαίως ε, είναι επένεται ε, η απλούστευση, αλλά απλούστευση δεν σημαίνει πάντα βελτίωση. Θα πρέπει βεβαίως να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε πως δεν θα χάσουμε χρήσιμους νομοθετικούς μηχανισμούς. Στα λιγότερο θετικά σημεία της έκθεσης, ο κύριος Λούτβιχσον βλέπει τρία σημεία κλειδιά που θα πρέπει να συζητηθούν πιο λεπτομερώς. Πρώτα απ' όλα έχουμε την αρχή ουδετερότητας των καυσίμων που θεωρεί προβληματική. Η αρχή αυτή αναφέρει πως όλα τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο στόχο πρέπει να φορολογούνται με το ίδιο ποσοστό. Ε, είναι λογική και δημιουργεί ένα ίσο πεδίο ανταγωνισμού, κάτι το οποίο βεβαίως μακροπρόθεσμα είναι λογικό. Κάθε καύσιμο έχει μια δίκαιη φορολογία, κάθε επενδυτική απόφαση θα βασίζεται σε μια προβλεψιμότητα. Υπάρχουν λογικές ανησυχίες της αυτοκινητοβιομηχανίας όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της αρχής, όσον αφορά το ντίζελ και την βενζίνη εφόσον οι στρατηγικοί τους έχουν ε, οικοδομηθεί γύρω από τις κινητήρες diesel, υπάρχει λόγος να είμαστε προσεκτικοί ε, στο τι θα γίνει στην πράξη στο πλαίσιο αυτό όμως δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε ε, όσον αφορά τον αντίκτυπο εφαρμογής αυτής της αρχής. Τα κράτη-μέλη δεν θα αλλάξουν τις, ε, τη σχέση αυτή μόνο με το να αυξήσουν την τιμή του ντίζελ. Ανταυτού, οι περισσότερες εθνικές στρατηγικές μάλλον θα πάνε σε ένα συνδυασμό μείωσης φορολογίας βενζίνης και αύξησης φορολογίας του ντίζελ. Η λύση εδώ πέρα θα πρέπει να ε, λάβει υπόψη βεβαίω και την καταληκτική ημερομηνία του 2023 για τα καύσιμα κινητήρων και θα πρέπει να υπάρχει μια σταδιακή μετάβαση προς την ουδετερότητα ξεκινώντας από το 2023 και θα πρέπει να οδηγηθούν μέχρι τότε τα κράτη-μέλη στην ουδετερότητα. Και άρα μέσω ενός λογικού μηχανισμού θα έχουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τις αυτοκινητομηχανίες για να μπορέσουν να προσαρμοστούν λογικά. Η λύση άρα δεν είναι να καταργηθεί η αρχή της ουδετερότητας των καυσίμων, καθώς δεν υπάρχουν ουσιαστικές δυσκολίες που να προβλέπονται σε κανέναν άλλο τομέα, δεν υπάρχουν άρα πιστικά επιχειρήματα για να καταργηθεί η αρχή αυτή. Το δεύτερο είναι το ότι ανισχύει η κυρία Λούλινγκ για την αυτόματη αναπροσαρμογή των ελάχιστων φορολογικών ε, επιπέδων και πως αυτό θα δημιουργήσει πληθωρισμό. Είναι δικαιολογημένη αυτή η ανισχύα, μόνο εάν ε, επιλεχθεί ένα ποσοστό το οποίο δεν είναι σωστό. Εφόσον η Κομισιόν αντιθέτως επέλεξε ένα κατάλληλο ποσοστό το οποίο εξαιρεί τα προϊόντα ενέργειας, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε πως η τιμαριθμική αναπροσαρμογή θα δημιουργήσει πληθωρισμό. Για να πάμε και στον πραγματικό κόσμο, η Σουηδία έχει ευθυγραμμίσει τις ε, φορολογίες και διοξιδίου του άνθρακα και ενεργειακού περιεχομένου με τις τιμές καταναλωτών χωρί να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα πληθωρισμού. Οπότε θα πρέπει να γίνει αυτό για να μην καταλήξουμε στο να μην σημαίνουν τίποτα αυτά τα επίπεδα. το 2003, στο πλαίσιο αυτής τη οδηγία πάρα πολλά μέτρα έχουν καταστεί ανενεργά και θα πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτή τη δυναμική. Τρίτο και τελευταίο, Υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν ανανεώσιμα καύσιμα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς στο σχέδιο έκθεσης στην πρόταση Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει δουλειά για να επιτύχουμε τα πράγματα σωστά εδώ πέρα. Σε... Επιπλέον, πέρα από αυτά τα οποία αναφέρονται στο σχέδιο έκθεση πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένε πτυχέ. Πρώτον, λογικό θα είναι οι υποχρεωτικέ φοροαπαλλαγές ε, στον τομέα των αμεταφόρων και των θαλασσίων μεταφορών να γίνουν προαιρετικέ ε, καθώ οι απαγορεύσει από πλευρά, επικουρικότητα δημιουργούν προβλήματα και δεν ε, έχουν τη βάση του σε διεθνή νομοθεσία. Δεύτερον, τωρινή δυνατότητα απαλλαγή των καυσίμων για τροφίμων Νοικοκυριό, με συγχωρείτε, θα πρέπει να επανεξεταστεί, καθώς θα πρέπει να δοθεί ένα κίνητρο επενδύσεις ε, σε ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Τρίτον, ενδιαφέρον θα είναι να προωθηθεί η εισαγωγή υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων μέσω μιας προσωρινής απαλλαγής ε, του ηλεκτρισμού αυτών των οχημάτων. Και τελευταίο, η ιδέα της Κομισιόν του να μην αντιμετωπιστούν κάποια ζητήματα παρά μόνο μετά το 2015 είναι κάτι το επιμαχώ. Όλες οι αποφάσεις αρχής πρέπει να ληφθούν τώρα και μετά οι τεχνικές ρυθμίσεις να γίνουν από την Κομισιόν από το 2015 και μετά. Αλλιώς υπάρχει ένας κίνδυνος να μπλοκαριστούν αποφάσεις οι οποίες έχουν ζωτική σημασία για να λειτουργήσει σωστά η οδηγία. Συνοψίζοντας λοιπόν το σχέδιο έκθεση είναι μια πάρα πολύ καλή βάση συζητήσεων του επόμενου εβδομάδες και μήνες. Okay, thank you very much. Uh, next for... Ευχαριστώ πολύ, Φίλιπ Ντιμπάλκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λουλίνγκ για το σχέδιο έκθεσης και για τη συνεργασία. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες γενικές αρχές που θα πρέπει να έχουμε υπόψη όσον αφορά την κατάθεση κάποιων τροπολογιών. Θεωρώ πως είναι αυτή η οδηγία φορολόγησης ε, της ε, ενέργειας δεν ε, έχει πουθενά ως ε, στόχο την αύξηση της φορολογίας. Αυτό αφορά μόνο δημοσιονομικούς ε, στόχους και δικαίως βεβαίως τα αναφέρει αυτά η κυρία Λούλινγκ. Και μια δεύτερη γενική αρχή που θα ήθελα να αναφέρω είναι πως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ίδιες, ίσες συνθήκες ανταγωνισμού όσον αφορά όλες τις μορφές ενέργειας και συμφωνώ επίσης με την διπλή αυτή ε, φορολόγηση και του διοξιδίου του άνθρακα και του, της περιεκτικότητας σε ενέργεια και όσον αφορά βεβαίως και τους καταναλωτές και τη βιομηχανία. Βεβαίω θα, θα πρέπει να επιτύχουμε και τους κλιματικούς ε, στόχους μας και βεβαίως ε, σας παραπέμπω εδώ πέρα στην λευκή βίβλο για τις μεταφορές που λέει ότι θα πρέπει να μειωθεί η εξάρτησή μας α, όσον αφορά την ενέργεια και οι εναλλακτικέ πηγέ ε, ενέργεια και θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβαστικό κείμενο. Ταυτόχρονα θεωρώ πω θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστικοί, αλλά βεβαίω και ε, φιλόδοξοι πρώτα απ' όλα ω ε, κοινοβούλιο και θα πρέπει να δούμε βεβαίως το πώς αντιμετωπίζει την αρχή τη επικουρικότητα η εισηγήτρια. Είναι σημαντικό βεβαίως να έχουμε και ίσες συνθήκες ανταγωνισμού. Δεν θα πρέπει να αποφασίζει το κράτος ποια ε, πηγή ενέργειας θα χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να είναι ίση φορολόγηση και να μπορέσει να αποφασίσει η αγορά. Τώρα, με ποιο βαθμό μπορεί να επιτευχθεί αυτή η επικουρικότητα δεν θεωρώ πως θα πρέπει να γίνει ε, οπωσδήποτε μέσω του να ανέβει η τιμή του ντίζελ, αλλά θα μπορούσε να πέσει και λίγο η τιμή της βενζίνης. Όπως γίνεται σε κάποια κράτη-μέλη. Ναι, επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος για να δοθεί χρόνος και στον καταναλωτή και στη βιομηχανία να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση καθώς υπάρχουν και επενδυτικοί κύκλοι της βιομηχανίας που βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντική. Είδα κάποια στατιστικά στοιχεία που λένε πως η αύξηση της τιμής του δίζελ δεν θα έχει άμεση επίπτωση στον αριθμό αυτοκινήτων δίζελ που θα πολλούνται. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Αλλού συμφωνώ με την εισηγήτρια αυτόματη τη αριθμική αναπροσαρμογή είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει αντίθετους και είναι νομίζω κάτι ε, το απαράδεκτο. Δεν μπορεί τα ευρωπαϊκά ελάχιστα να τα προσαρμόζουμε αυτομάτως. Δεν γίνεται εξάλλου. Όπως ξέρετε, μαριθμική αναπροσαρμογή πλέον στους μισθούς. Δεν νομίζω λοιπόν να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στην ε, αριθμική αναπροσαρμογή των φόρων, την αυτόματη και των εσόδων του κράτους. Επίσης, για την εξαίρεση των οικοκυριών για κοινωνικούς λόγους. Ακριβώς θα πρέπει να δώσουμε και εδώ πέρα ένα μήνυμα για να μπορέσουν να αλλάξουν και τα νοικοκυριά την ε, συμπεριφορά τους ε, την ενεργειακή. Τέλος, για τομείς ε, έντασης ενέργειας δεν θα πρέπει να υπάρξει εδώ πέρα διπλή φορολογία και από το ETS και από αυτό εδώ το σύστημα. Νομίζω πως θα πρέπει να έχουν επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν και να υπάρξει βεβαίως ε, και η σχέση με τον τομέα, τον εθελοντικό τέλος. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημαντικά σημεία με τα οποία συμφωνούμε με την εισηγήτρια και τους υπόλοιπους σκιοδησηγητές και βεβαίως αναμένουμε το πώς θα μπορέσουμε να αναζητήσουμε συμβιβασμούς και είναι ένας πάρα πολύ πολύπλοκος φάκελος και νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε αρκετά φιλόδοξοι για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που θα μπορέσουμε να έχουμε το Συμβουλίο. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θυμάμαι, τέλη Αυγούστου είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και τότε εγώ είχα πει ότι θα ήθελα να συνεργαστώ με την κυρία Λούλινγκ και πρέπει να σας πω ότι είχα δίκιο τότε. Σας το λέω τώρα πια γιατί η κυρία Λούλη οργάνωσε ε, κάποιες ενδιαφέρουσες συναντήσεις, ε, κάποια σημαντικ, κάποιες σημαντικές ακροάσεις ε, για τα θέματα αυτά που αφορούν πολύ σημαντική νομοθεσία. Όμως, πάνω απ' όλα, θα ήθελα να την ευχαριστήσω γιατί έλαβε υπόψη της όλα τα ε, σημεία τα οποία θέλαμε να τις υποβάλουμε. Μερικές παρατηρήσεις εισαγωγικές. Λαμβάνοντας υπόψη την ε, συνολική συζήτηση, ε, θα ήθελα τελικά να αναφερθώ μονάχα στα πιο σημαντικά σημεία τα οποία αναφέρονται στην έκθεση αυτή. Πρώτον, η αρχή της αναλογικότητας. Σημερίζομαι απόλυτα την θέση της κυρίας Λούλινγκ. και εμείς ε, σαν ε, συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές ε, θα ζητήσουμε να καταργηθεί αυτή η αρχή της αναλογικότητας. Δεύτερον, αυτόματη μαριθμική αναπροσαρμογή των ελαχίστων τιμών. Και εδώ είμαστε κατά. Και αν κατάλαβα καλά και σε αυτή την περίπτωση έχουμε ίδια άποψη με την κυρία Λούλινγκ εξαιρέσεις για τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. Η συζήτηση αφορά ε, για το κατά πόσον αυτή η έκπτωση, αυτή η εξαίρεση μάλλον θα είναι ε, εθελοντική ή υποχρεωτική. Εμείς στηρίζουμε την εθελοντική θέση. Τελευταίο σημείο. Μεταβατική περίοδος. λαμβάνουμε τις μεταβατικές περιόδους πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Θεωρούμε ότι αυτές οι μεταβατικές περίοδοι είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει να δώσουν το χρόνο στην βιομηχανία έτσι ώστε να προσαρμοστεί και να προσαρμοστούν βεβαίως και οι καταναλωτές. Λοιπόν, νομίζω ότι στα περισσότερα σημεία της έκθεσης αυτής θα βρισκόμαστε πολύ κοντά στη θέση της κυρίας Λούλινγκ. Η κυρία Λούλινγκ στο τέλος αναφέρθηκε σε κάτι καινούριο, δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορες φήμες, ε, φήμες οι οποίες ε, αναφέρονται σε μια διαφορετική στάση του Συμβουλίου. Θα περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα, την τελική έκβαση των συζητήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ε, θα μιλήσει για το εξ του Φιλίπ. Ναι, εξ ε, του σκιώδους συζητή του της ομάδας μας Φίλιπ Λάμπερτ να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτον, να θυμίσω ότι εδώ ε, ασχολούμαστε με, τη, με τα οικονομικά ζητήματα και στο Πανεπιστήμιο μου μάθανε ότι η οικονομία ε, ισούται με την αποτελεσματικότητα. Ε, θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε θα πρέπει ε, να ε, δούμε την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος ενώ εδώ μιλάμε περισσότερο για την ε, μέσο πρόθεσμη, βρέχη πρόθεσμη αντίδραση της βιομηχανίας. Τώρα, εάν θέλουμε να κάνουμε ε, μακροπρόθεσμη φορολογική πολιτική, τότε ε, μπορούμε όντως να πούμε ότι μακροπρόθεσμα ε, το ντίζελ, ας πούμε, θα είναι αυτό το οποίο θα ευνοηθεί περισσότερο. Αλλά στο, στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου μίλησαν οι εκπρόσωποι της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας και αναφέρθηκαν σε ένα μοντέλο το οποίο δεν προσαρμόζεται στις κλιματικές αλλαγές. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα πρέπει τα συστήματα φορολόγησης της ενέργειας στον τομέα των καυσίμων θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και λογικά, δηλαδή θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και την ένταση χρήσης ενέργειας αλλά και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και, όπως, και επομένως θα πρέπει να είναι λογικά. Θα ήθελα να μου πει η συγγήτρια ε, ποια είναι η θέση της όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή την οικονομική αποτελεσματικότητα εάν ε, διαγραφεί αυτό το κομμάτι της προτάσεως. Επίσης πιστεύω ότι για να ε, κρατηθεί έτσι μια σταθε... ένα σταθερό επίπεδο ε, άχθους φορολογικής φορολογικού βάρους όσον αφορά την φορολόγηση των ε, καυσίμων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όταν από την αρχή η φορολόγηση είναι χαμηλή υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην αύξησή της εκ των υστέρων και επίσης η χρήση μπορεί να ε, μειώνεται και το είδαμε ε, και στον τομέα των δασμών όπου δεν έχει καμία έννοια να διαγράψει κανείς τη λογική της αυτόματης αναπροσαρμογής. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό το σύστημα της αυτόματης της αναπροσαρμογής. Όσον αφορά την προσαρμογή των τιμών διοξιδίου του άνθρακος, εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να γίνει με μεταρρυθμίση, αλλά με, κατα... με πράξη κατεξουσιοδότηση και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε καλύτερα να αντιμετωπίσουμε τις πιεστικές ανάγκες της κλιματικής αλλαγής. Όσον αφορά τις απαγορεύσεις, εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει βάσει της οδηγίας να απαγορεύεται στα κράτη-μέλη να ε, επιβάλλουν φορολόγηση στις ε, θαλάσσιες μεταφορές ή στις αεροπορικές ε, μεταφορές. Επίσης δεν θα πρέπει να, θα πρέπει να διατηρήσουν τη δυνατότητα να φορολογήσουν περαιτέρω τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα πρέπει καταρχήν να υπεραμεινθούμε της αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποτελεί βάση του κειμένου, δηλαδή να έχουμε οικονομικά ε, βιώσιμη και αποτελεσματική ε, φορολόγηση με απότερο στόχο την ε, μείωση των ε, εκπομπών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Θα ζητήσω λοιπόν την Επιτροπή μας εδώ να λάβει υπόψη της ότι η κλιματική αλλαγή ε, και στο παρελθόν και τώρα θεωρείται σαν η μεγαλύτερη, η παταγωδέστερη αποτυχία που είχαμε όσον αφορά την αγορά και επομένως θα πρέπει να δούμε το μέλλον από την σκοπιά της οικονομικής Οικονομικής Επιτροπής, την οποία εδώ εκπροσωπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις ομιλητές έχω ακόμα εγγεγραμμένους. Αλλά έχω μόνο τρία, έξι λεπτά, συγγνώμη, θεωρητικά. Θα, ζητώ, λοιπόν, θα ζητήσω λοιπόν να κάνουν οικονομία χρόνου οι εισηγητές. Λάγεν, Hans-Peter Martin, Λάγεν. Μπορεί να μιλήσουμε όλοι και η Κομισιόν και εμείς. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Το θέμα δεν είναι αυτή τη στιγμή το ακριβές ύψος της φορολογίας. Οι προτάσεις Κομισιόν ακόμα και στις χώρες χαμηλής φορολογίας είναι κάτω από το υφιστάμενο ύψος των φόρων. Οπότε δεν υπάρχει πουθενά ε, υποχρέωση αύξηση των φόρων. Πρώτον. Δεύτερον, γίνεται διαρθρωτική πολιτική η οποία είναι αντίστοιχη με τις ε, μέχρι τώρα αποφάσεις κομισιών. Δεν το ξέρουν ε, πολλοί νέοι συνάδελφοι. Εγώ ήμουν ε, εισηγητής το 2008 για το διοξείδιο του άνθρακα των αυτοκινήτων και στην Επιτροπή Βιομηχανίας και ο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τότε εσκεμένα το τα νέα αυτοκίνητα τα είδαμε υπό το πρίσμα της μείωσης των εκπομπών. Και δεν συμφωνούσε τότε η Greenpeace και η Λυπή, αλλά το υπόλοιπο κοινοβούλιο το ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία. Οπότε ε, σκεμμένα προωθήσαμε τις ε, τεχνολογίες ε, μείωση χρήση τεχνολογία και δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανεί πω ο κινητήρα ο δίζελ σε σχέση με τον κανονική βενζίνη έχει σαφώς ε, χαμηλότερες εκπομπές και 89% των φορτηγών κινείται με ε, δίζελ. Και η πρόταση της Κομισιόν ήταν να φορολογηθούν όλα τα καύσιμα ε, με τον ίδιο τρόπο. Αλλά αν το κάναμε αυτό θα είχαμε αύξηση της τιμής του ντίζελ. Αυτή δεν θα ήταν περιβαλλοντική πολιτική, θα ήταν τεχνολογική πολιτική. Και στο παράδειγμα αυτό εδώ πέρα φαίνεται ακριβώς το λάθος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή η μία χείρα θέλει μείωση του διοξιδίου του άνθρακα το οποίο υποστηρίζουμε και η άλλη χείρα ταυτόχρονα στον ίδιο τομέα κάνει ακριβώς το αντίθετο. Όσο δεν υπάρχει μία ενιαία πολιτική και λογική στην Ευρωπαϊκή Κομισιόν δεν θα φύγουμε από το δίλημα του κατακρεματισμού των αρμοδιοτήτων. Γι' αυτό σας λέω πως δεν θα οδηγηθούμε αυτομάτως σε αύξηση της ε, φορολογίας γιατί όπως σας είπα αυτά το έχουν προτεθεί είναι κάτω από τους υφιστάμενους φόρους αλλά ε, έχουμε μια αναβολή των αποφάσεων που έχουμε λάβει είναι ζήτημα επικουρικότητας των κρατών μελών που εξακολουθούν να είναι υπεύθυνα για τη φορολογία και βεβαίως υπάρχει και η αρχή της ομοφωνίας. Και δεν είναι μόνο η Γερμανία όπως λέει ο κύριος Γκίγκολτ. Εξάλλου η Γερμανία τώρα ε, το έχει διαδώσει αυτό το θέμα, αλλά και οι χώρες όλες οι οποίες είναι υπέρ μιας λογική τέτοιας πολιτικής... είτε μιλάμε για την Γαλλία, την Ιταλία, είτε η Γερμανία, η Ολλανδία, δεν μπορούμε σε ένα δομικό ζήτημα να κάνουμε προτάσεις οι οποίες θα έχουν το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα από αυτό το οποίο θέλει η Κομισιόν και μετά να έχουμε τόσες πολλές εξαιρέσεις. Τις ανέφερε ο κύριος Σκυλούνα, ποιε ήταν ε, αυτό το οποίο κατέφεραν εκεί πέρα οι Βόροι. Γιατί τι έγινε. Ε, θα πρότεινε αυτά Επίτροπος Κλίματος και μετά τα, τα απέσυρε Δεν είναι λογική αυτή των σοσιαλδημοκρατών. Και καλά το λέει η κυρία Λούλινγκ, αλλά ε, θέλετε να πείτε κάτι στην κυρία Λούλινγκ. Δεν είναι, μην χρησιμοποιείτε την ιδεολογία. Και σας εγγυώμαι πως θα έχετε απέναντί σας την πλειοψηφία των Υπουργών, γιατί δεν είναι λογική αυτή η προσέγγιση και δεν ακολουθεί η Κομισιόν αυτά τα οποία προτείνει αλλού άλλη υπηρεσία της. Ευχαριστώ, Ρομπέρ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όπως ξέρουμε, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με αγαθές προθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση οδηγίες που χαρακτηρίζεται αυτό το φιλοπεριβαλλοντικό ε, αγγελικό προσανατολισμό που συνοψίζεται στο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σώσει από μόνη της ολόκληρο τον πλανήτη». Φαίνεται ότι στόχος οδηγίας είναι να φορολογήσει, να φορολογεί και να φορολογεί συνέχεια. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει και ένα σύστημα αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των φόρων. Όταν μας λένε λοιπόν ότι μέχρι το 2020 θα έχουμε 20 δισεκατομμύρια περισσότερα φορολογικά έσοδα. Φυσικά αυτό θα χαροποιήσει τους Υπουργούς Οικονομικών. Αλλά αυτό θα επηρεάσει το πορτοφόλι των ε, συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των πιο χαμηλών εισοδημάτων που δεν μπορούν ε, να στερηθούν και το γιοταχή τους. Και 20 δισεκατομμύρια επιπλέον φορολογικά έσοδα δεν θα είναι το τέλος του δρόμου, γιατί όλα αυτά θα τύχουν και κάποια στιγμή αριθμική αναπροσαρμογή με την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, αύξηση του πληθωρισμού. Παράλληλα στι διαβεβαιώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η αύξηση θα οδηγήσει και σε αύξηση του πληθωρισμού. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με του οικονομικού μα στόχου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρώτα απ' όλα, πάνω απ' όλα, η οδηγία αυτή θα πλήξει τα εκατομμύρια αυτοκινητιστών που αγόρασαν αυτοκίνητα με κινητήρες δίζελ. Γιατί όλοι συμφωνούμε ότι οι κινητήρες δίζελ είναι πιο, αποτελεσ... πιο οικονομικοί από τους κινητήρες που, και, που Αυτό ισχύει. Αλλά με τα νέα μέτρα θα πληγούν και αυτοί οι αγοραστές, οι καταναλωτές. Και φυσικά το λόμπι, το πετρελαϊκό, επικροτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Και αυτό που με εκπλήσει είναι ότι συμφωνούν με το πετρελαϊκό λόμπι και οι πράσινοι. Γιατί η παραγωγή βενζίνης και δίζελ έχουν προβλήματα. Γιατί ο κόσμος διάλεξε ε, μαζικά τα, τους κινητήρες δίζελ και άρα δεν υπάρχει ζήτηση αρκετή για βενζίνη. Εξού και το ενδιαφέρον του πετρελαϊκού λόμπι για την οδηγία. Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να υποταχθώ στη λογική αυτή. Θα υποβάλω λοιπόν τροπολογία ζητώντας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίψει Α, δύο μάλιστα θα υποβάλουμε τη σχετική οδηγία, να υπορρίψει ε, σύλληδιν αυτή την πρόταση οδηγίας. Και αν δεν εγκριθεί η τροπολογία αυτή, θα συνταχθώ με τις προτάσεις ε, της εισηγητριάς μας. Και ευελπιστώ ότι το Συμβούλιο ε, θα ε, καταρρύψει αυτή την οδηγία θα οδηγεί σε έκτρωση αυτή τη οδηγία. Εγώ ήμουν ανέκαθεν υπέρ του δικαιώματο σε άμβλωση. Ελπίζω να ισχύσει άμβλωση και για την οδηγία αυτή. Ευχαριστώ. Έχουμε ξεπεράσει ήδη το ωράριό μα για αυτή τη συζήτηση. Δεν θα ήθελα να διακοθεί περαιτέρω ο κατάλογο των ομιλητών. Ο Χάν Πίτερ Μάρτιν. Ευχαριστώ. Ω υποστηρικτή του Diesel, ξέρετε, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Για τα λόμπι μπορώ. Δεν το εννοούσα έτσι κύριε Λάγκεν, Πάντα ο κύριος Μάρτιν σε σχόλιο εκτός μικροφώνου. Για τα λόμπι τώρα και τους πράσινους ε, υπάρχουν και άλλα λόμπι, υπάρχει και το λόμπι της ατομικής ενέργειας και εδώ πέρα κυρία Λούλινγκ ε, υπάρχει, υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις που με ενοχλούν π.χ. στην τροπολογία 1 μιλάτε για στόχους βιομηχανικής πολιτικής ε, και μετά παρακάτω μιλάτε για την διαγραφή της ενέργειας ε, από ανανεώσιμες πηγές, οπότε βλέπετε από ποια οπτική σκοπιά ε, το έχετε γράψει. Οπωσδήποτε υπάρχει μια θεμελιώδης ε, οικονομική συζήτηση για την αυτόματη μεριθμική αναπροσαρμογή των φόρων και το τι πληθωρισμό θα προκαλέσει, αλλά βεβαίως μην ξεχνάμε πως υπάρχει αυτό το οποίο λέτε εσείς πάντα, το να υπάρχει μια προβλεψιμότητα της εξέλιξης των τιμών. Κλασικό παράδειγμα βεβαίως είναι εδώ πέρα οι καταλήτες, όπου μας λέγατε για το όνομα του Θεού θα καταστραφεί η αυτοκινητομηχανία κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε και ξέρετε πως ε, αυτά τα οποία έγιναν τότε δεν ε, ωφέλησαν μόνο το Λος Άντζελες και τη μείωση του νέφους αλλά και την μηχανία Και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να μην υπάρχει ένα ντάμπινγκ τιμών στον τομέα της φορολόγησης της ενέργειας αλλά να υπάρχει μια α, αξιόπιστη, μια λογική αναπροσαρμογή και βεβαίως ε, να μην μιλάμε μόνο για το κλίμα, αλλά να κάνουμε κάτι και στον τομέα των τιμών. Και ε, πολλοί λένε βεβαίω πω είναι σημαντικό το ζήτημα του κλίματο, θα πρέπει να θεωρήσουν οι ίδιοι άρα πω και η δημαριθμική αναπροσαρμογή είναι εξίσου σημαντική. Ευχαριστώ πολύ. Είπα ήδη ότι η Κομισιόν δεν θα μιλήσει. Άσε, θε να πει κάτι πολύ σύντομα. Όχι. Όχι, κυρία Πρόεδρε, λέει η κυρία Λούλινγκ. οφείλω να διαπιστώσω ότι η σοσιαλιστική ομάδα έχει δύο ακραίες θέσεις. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου, ότι κρίμα λέει η κυρία Λούλινγκ. Θα πρέπει να πείσεις την ομάδα σου. Α, κοίτα αν αυτό ισχύει που μου λες, οι διερμηνείς δεν το άκουσαν, ε, τότε θα πρέπει να διαπιστώσω ότι από τη στιγμή που η ομάδα μου είναι μαζί μου, τότε παραμένει ένα κομμάτι που δεν έχει καθόλου γνώμη, δεν έχει καθόλου άποψη. Τι να κάνω, να βασιστώ και σε αυτούς για να επιτύχω την πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει. Αυτά που είπε ο εισηγητής ε, των ε, φιλελεύθερων, ε, είναι πολύ ενδιαφέροντα, τον, τον ευχαριστώ. Ο σκιώδης συγητής ε, των ε, συντηρητικών μεταρρυθμιστών με στήριξε πολύ, τον ευχαριστώ, αλλά Νομίζω ότι πρέπει να διορθώσουμε εδώ ότι έγινε ένα λάθος, δηλαδή ότι η ομάδα ECR είναι ε, ε, υπέρ της υποχρεωτικής έκπτωσης του φόρου για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, όχι δηλαδή σε εθελοντική βάση. Έκανε λάθος ο εισηγητής προηγουμένως όταν το ανέφερε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά κυρία Πρόεδρε και θα προσπαθήσω να βρω πλειοψηφία που θα στηρίξει την ε, ε, έκθεσή μου. Αλλά για την ώρα και από αυτά που άκουσα δεν μπορώ να εξάγω πολύ σαφή συμπεράσματα, κυρίως γιατί η σοσιαλιστική ομάδα είναι χωρισμένη αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να βρεθεί λοιπόν εκεί η συνένεση επί συγκεκριμένης ε, γνώμης, ε, μια γνωμοδότηση βεβαίως και μια άποψη την οποία δεν θα ρίξω Συμβούλιο απευθείας στον κάλαθο των αχρήστων. Ωραία, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 16η Νοεμβρίου στις 6 ε, το απόγευμα. Θα συζητηθούν οι τροπολογίες στα 9 Δεκεμβρίου, θα ψηφίσουμε στις 24 Ιανουαρίου στην έκθεσή μας και στην Ολομέλεια, ε, θα συζητηθεί την πρώτη Ολομέλεια του Μαρτίου. Ε, θα δούμε τι θα γίνει και με το Συμβούλιο. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε. Θα δούμε, μπορούμε να καθυστερήσουμε την έκθεσή μας, θα δούμε πώς θα έχει, θα βολιδοσκοπήσουμε λίγο την κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε επίσης, λέει η κυρία Λούλινγκ, πότε μπορούμε να έχουμε τις γνωμοδοτήσεις από τις διάφορες επιτροπές, γιατί καλό θα ήταν να ξέρουμε πότε θα είναι σε θέση να εγκρίνουν οι διάφορες επιτροπές τις γνωμοδοτήσεις τους, ε, γιατί βλέπω ότι οι γνωμοδοτήσεις ε, είναι πολύ ακραίες, φτάνουν από τη μία άκρη στην άλλη και επομένως ενδεχομένως θα υπάρχουν και πολλές ε, ε, τροπολογίες θα δούμε. Ναι, ναι, πρέπει να έχεις και χρόνο να τις συζητήσεις. Ε, θα δούμε λοιπόν. Εμείς θα προσπαθήσουμε πάντως να είμαστε πιο ευέλικτοι. Βέρνερ. Μια σύντομη παρατήρηση πως εδώ πέρα υπήρχε διαφωνία με την ε, Επιτροπή Βιομηχανίας για το εάν η λύση ήταν η στενή συνεργασία και θα πρέπει τουλάχιστον να περιμένουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας. Αυτή ήταν η λύση. Θα προσπαθήσουμε να περιμένουμε τις γνωμοδοτήσεις τους και να έχουμε και το χρόνο να το καλοσκεφτούμε πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Θα περάσουμε τώρα στο σημείο 6, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού των Οικονομικών Πολιτικών. Η συγκίτρια είναι υπερβάως. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ το σύνολο των συναδέλφων που δέχτηκαν να ξανανοίξει το θέμα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την επικαιρότητα η οποία κάθε μέρα δίνει και συμπληρωματικά στοιχεία. Κόπτια Je dois dire que j'ai été un peu surpris πρέπει να πω ότι εξεπλάγει λίγο από τον Προεδρεύοντα του ΕΚΟΦΗΝ ε, γιατί όταν ε, προσπάθησα να καταλάβω τι γίνεται ε, μου είπε ότι δεν αναφέρεται στα συμπεράσματα του ε, Συμβουλίου σε αυτό το Europlus, αλλά εγώ ε, το βλέπω να αναφέρεται τουλάχιστον τρεις φορές. Εν πάση περιπτώσει, ίσως διαβάζουμε διαφορετικά τα συμπεράσματα. Θα ήθελα να επιμείνω επί πέντε σημείων, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Πρώτο, όπως το παρουσιάζει σήμερα η Επιτροπή τα πράγματα, έχουμε την εντύπωση ότι είναι μία ακόμα διαδικασία, μία ακόμα γραφειοκρατική κίνηση και όχι ένα σημαντικό εργαλείο πολιτικής όπως θα όφιλε να είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ε, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτή η ε, ετήσια αναθεώρηση της ε, ανάπτυξης είναι ή θα όφιλε να είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο και ε, οπωσδήποτε το σχέδιο Europlus θα πρέπει να ε, ενσωματωθεί σε αυτήν την αξιολόγηση. Δεν είναι δυνατόν να ηγούμεθα μιας ε, τέτοιας άσκησης, μιας, ενός ευρωπαϊκού εξαμήνου, εάν δεν έχουμε και κάποιο συγκεκριμένο προσανατολισμό ετήσιο όσον αφορά την ανάπτυξη. Τώρα και αν βεβαίως τις βάλουμε και επιθετικό προσανατολισμό, προσδιορισμό, να είναι αηφόρος, να είναι βιώσιμη, θα είναι ακόμα καλύτερα. Δεύτερο σημαντικό κατά την άποψή μου σημείο, ο τρόπος με τον οποίο ε, χειριζόμαστε την ε, παλαιά παράγραφο 30 του ψηφίσματος, εκεί δηλαδή που εγώ πρότεινα την δημιουργία ειδική υποεπιτροπής για την Ευρωζώνη. Μπερδεύεται ακόμα περισσότερο η πρόταση αυτή, την οποία πολλοί θεώρησαν προκλητική. Ξέρετε ότι ξεκίνησα μια επιστολογραφία ε, με τους συναδέλφους, με τον συνάδελφο μάλλον της ε, ΑΦΚΟ και προτείναμε με τον ε, σκιώδη Σιγητή ε, μια συμβιβαστική τροπολογία όπου λέμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξελίσσει τις ε, δομές του με αυτές του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Βεβαίως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής ε, της Ευρωζώνης οι συνθήκες αλλάζουν και μάλιστα προχωρούν οι διαρθρώσεις τελείως διαφορετικά και μόλις είπατε μάλιστα και ότι ο νέος, ε, ε, ο νέος επίτροπος στις 23 Νοεμβρίου θα υποστεί μια νέα ακρόαση βάσει των νέων του αρμοδιοτήτων. Πότε λοιπόν θα αποφασίσει και το Κοινοβούλιο ότι θα μπορεί ή θα οφείλει ε, να προσαρμόσει τις δομές του. Πάντως η πρόταση που είχα κάνει δεν είναι πρόταση ε, για διχασμό του Κοινοβουλίου. Είναι μία πρόταση σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να δούμε τον παραλληλισμό των εξουσιών ε, και την ε, προώθηση της δημοκρατικής λογοδοσίας γιατί διαφορετικά εγώ φοβάμαι ότι τα πράγματα θα λαμβάνουν χώρα στα εθνικά κοινοβούλια και ότι εμείς δεν θα έχουμε καθόλου χώρο για ευρωπαϊκή συζήτηση. Τρίτον, ο τρόπος ε, συνεταιρισμού ή συνεργασίας με τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου με τον οποίο ε, οποίων ε, ε, έχουμε οργανώσει την ε, συνάντηση του επομένου Φεβρουαρίου ανάμεσα στην Οικονομική Επιτροπή και, τις, και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Νομίζω ότι ακολουθούμε τον ευκταίο δρόμο. Τέταρτο σημείο το οποίο ήθελα να αναφέρω είναι η φύση της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εδώ προκύπτει το ερώτημα. Ζητούμε συν απόφαση για το Κοινοβούλιο, δικαίωμα συν απόφαση για το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι εάν θέλουμε να είμαστε συνεκτικοί, οπωσδήποτε θα πρέπει να περάσουμε από αυτή τη συζήτηση για τη συναπόφαση. Το, ας πούμε, ε, είμαστε συνομοθέτες στο Six Pack ή στο καινούριο άρθρο 136. Ωραία. Αλλά η ουσιώδης πράξη, η πράξη πράξη ε, για, την, ε, την οικονομική πολιτική είναι η συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Σε κάθε δημοκρατία έτσι συμβαίνει. Εδώ και υπερβολικά πολύ καιρό γίνεται λόγος για αυτό το θέμα. Όταν συζητούσαμε για τη στρατηγική της Λισαβόνας, ε, λέγαμε ότι εντάξει, ας υπάρχει μία πρόταση μετά από πρωτοβουλία των ομάδων εν ώψη των συμβουλίων, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Αφιερώνουμε χρόνο και χρήμα για ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι μηδαμινό το τονίζω, είναι μηδαμινό. Αυτό θα πρέπει να ξαναδούμε. Αυτό το κοινοβούλιο λέει κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβει υπόψη το Συμβούλιο όσον αφορά τους οικονομικούς προσανατολισμούς δεν λέω ότι με την παρούσα πλειοψηφία του Κοινοβουλίου οι επιλεγμένοι, οι αποφασισμένοι οικονομικοί προσανατολισμοί θα μου άρεσαν πάντοτε, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα, να δείξουμε κάτι απέναντι στο Συμβούλιο. Και επίσης ε, η συναπόφαση λέει δεν λειτουργεί σε τρεις μήνες. Ναι, αλλά θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Θα πρέπει να βρούμε και το χρόνο και τα μέσα έτσι ώστε ε, γενικά πολλό δε μάλλον περισσότερο που προφανώς τέλη Νοεμβρίου η Κομισιόν θα βάλει και καινούργια στοιχεία στο τραπέζι. Μέχρι, λοιπόν, από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει δυνατότητα συναπόφασης για τους μεγάλους οικονομικούς προσανατολισμούς, για το, για το ευρωπαϊκό εξάμεινο όπως θέλετε πέστε το. Γιατί αν συνεχίσουμε να λέμε στο Συμβούλιο ή στην Κομισιόν, ε, ξέρετε πρέπει να λαμβάνετε και υπόψη σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα πάμε πουθενά, δεν θα προχωρήσουμε. Τελευταίο συζητήθηκαν κάποια πράγματα στο Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα ε, και στο, στη Σύνοδο της ε, Τετάρτης. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καμία εντολή από την ομάδα μου για να πω οτιδήποτε. Εγώ το λέω γιατί το σκέφτομαι και θέλω να το συζητήσουμε μεταξύ μας. Νομίζω ότι στο Συμβούλιο κάποιες χώρες, όχι οι πιο αδύναμες, θέλουν αναθεώρηση της συνθήκης και θέλουν την αναθεώρηση πώς το γράφει να δείτε στα συμπεράσματα. Ε, θέλουν λοιπόν να κάνουν περιορισμένες τροποποιήσεις ε, των, των συνθήκων. μοντιφικασιών λιμιτές, στα γαλλικά. Και έχω την εντύπωση ότι τελικά περίμενα να, πούν, να πούμε αυτό που ανεμένετο να πούμε. Εγώ νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί έστω και αν ε, λαμβάνοντα υπόψη την ε, πολιτική κατάσταση στη χώρα που θα προτιμούσε η συζήτηση αυτή να μην ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου. Παρόλα αυτά λέω ότι το, Κοινοβούλιο θα πρέπει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προετοιμαστεί για αυτή τη συζήτηση γιατί διαφορετικά στο Συμβούλιο κάποιες χώρες ε, θα αποφασίσουν και θα πούν ποια θα είναι η τροποποίηση των συνθήκων και τι θα αφορά. Επομένως εγώ λέω ότι θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει γύρω από μια οικονομική πολιτική η οποία θα του διασφαλίσει και την αλληλεγγύη και την ε, δημοκρατία και την ανταγωνιστικότητα. Επομένως επιλέγουμε είτε να μην κάνουμε τίποτα και θα περιμένουμε λοιπόν τον οδικό χάρτη του Συμβουλίου ή θα αποφασίσουμε να κινηθούμε έγκαιρα και πρόημα ε, και επομένως να βγούμε μπροστά από το Συμβούλιο. Αυτά ήταν τα λίγα στοιχεία τα οποία ήθελα να πω έτσι ώστε να δώσω, ρίξω λίγο φως σε αυτή τη συμβαστική λύση που προτείνω. Ξέρω ότι στα πλαίσια της Επιτροπής μας εδώ υπάρχει μια γραμμή συνένεσης η οποία λέει ότι το ε, six-pack και μόνο αυτό. Συμφωνώ ότι αυτό το εξάπτυχο, ας πούμε, αυτή η εξάπτυχη ε, δέσμη είναι κάτι θετικό, αλλά αυτό ήταν στην αρχή. Και αν διαβάσετε όμως προσεκτικά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, αναφέρεται ρητά στην παράγραφο 5 σημαντική ενδυνάμωση του συντονισμού και της εποπτείας σε δημοσιονομικό και οικονομικό επίπεδο με τρόπο συγκεκριμένο που θα ξεπερνάει το πακέτο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση ε, και αυτό θα εφαρμοστεί ε, γρήγορα και επομένως εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε με προσοχή αυτό το συμπέρασμα της Συνόδου ε, Κορυφής γιατί εάν δεν αναγνώσουμε προσεκτικά τα συμπεράσματα τότε θα μας προσπεράσουν οι καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ζαν Πολ Γκόζες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αν θέλουμε να χρησιμεύσει κάτι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν θέλουμε να είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό, θα πρέπει να είναι διορατικό, να προλαμβάνει τις εξελίξεις. Εγώ κάθε φορά που, που έχω επαφή με πολίτες, με δημοσιογράφους, με ρωτά συνέχεια και όλοι το ίδιο. Τι κάνει επιτέλους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσφατα είχα και μια συνέντευξη την περασμένη Παρασκευή στο, στη Φράση Info. Όλοι αυτοί με ρωτάνε, μα τι κάνει επιτέλους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω ε, την αίσθηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, προσπαθεί να κρατήσει τη συνείδησή του εγκρίνοντας εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις, ψηφίσματα που δεν ξέρουν και πολλοί σε τι χρησιμεύουν. Αυτή τη στιγμή όλοι αναγνωρίζουμε το δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει και όσοι είναι κατά της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα του δημοκρατικού ελλείμματος και βάλλονται κατά του κοινοβουλίου. Δεν είναι όμως το κοινοβούλιο που χαρακτηρίζεται αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα. Ίσα ίσα έχει δημοκρατική νομοποίηση πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε θεσμικό όργανο. Το δημοκρατικό έλλειμμα οφείλεται στο γεγονό ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται και αυτές που αφήνουν στίγμα στην κοινή γνώμη και οι πιο σημαντικές λαμβάνονται από τους κυβερνώντες που φυσικά έχουν απορρεύσει από την λαϊκή ετοιμιγορία αλλά όχι άμεσα. Οπότε νομίζω ότι είναι πραγματικά... Ε, έχει φτάσει το κόμπο στο χτένι να ξεφύγουμε από την πεπατημένη, να ξεφύγουμε από, την, ε, από το καθυσυχασμό, φυσικασμό της συνείδησης που μας έχει χαρακτηρίσει μέχρι τώρα. Οπότε, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, δύο είναι οι προσανατολισμοί, όπως λέει η έκθεση. Τι θα πρέπει να κάνουμε στα τρέχοντα και δεύτερον, τι θα πρέπει να τροποποιήσουμε προκειμένου να δώσουμε μια πιο ισχυρή δημοκρατική βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια της εισηγητρίας, η Υποεπιτροπή ξέρω ότι τουλάχιστον θεωρούμε στην ομάδα μου ότι αυτά που έκανε δεν είναι αρκετά και ε, οι περισσότερες χώρες ε, που είναι εκτός Ευρωζώνης, εκτός από δύο, κάποια στιγμή θα μπουν στην Ευρωζώνη, οπότε ενδιαφέρονται από τα μέτρα που θα ληφθούν στον τομέα αυτό. Πάντως είναι λογικό να λάβουμε υπόψη και τις εξελίξεις ε, στις κυβερνήσεις ε, ε, σε τη φορά ιδιαίτερα την οργάνωση της Ευρωζώνης. Και ίσως αν έχουμε μία οργάνωση καθρέφτη που θα αντανακλά αυτά που γίνονται στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρήσιμη. Αλλά φυσικά αυτή θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί. Άλλο σημαντικό θέμα αυτό τη συναπόφασης. Για το ζήτημα αυτό, οι πρωταρχικές μου παρατηρήσεις ε, θα τάσσονταν υπέρ τη συμπερίληψη τη συναπόφασης στου προσανατολισμούς τη οικονομική πολιτική. Με ποιο όμω τρόπο, με ρεαλιστικό τρόπο. Μιλήσαμε για προθεσμίε και είναι πολύ σημαντικό να μην ε, χαθούμε σε ατέρμονες συζητήσεις που θα αποδυναμώσουν ουσιαστικά τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάτι άλλο που θα πρέπει να αποφύγουμε είναι να επισέλθουμε ε, σε υπερβολικά σχολαστικές λεπτομέρειες που είναι ε, και περιτές και δεν είναι και ρεαλιστικέ και δεν εξυπηρετούν το πνεύμα της καλύτερου, του καλύτερου οικονομικού συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε σημαντικέ αναλύσει, να επιδείξουμε ευρηματικότητα, φαντασία, δημιουργικότητα. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό στην έκθεση αυτή να γίνεται μνήα και της αναζήτησης μεθόδων συναπόφασης. Ίσως το Κοινοβούλιο δεν θα υποβάλει τη θαυματουργή λύση, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε κάποιες κατεπίγουσες διαδικασίες με αμοιβαία συνεννόηση και κατανόηση, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στο Κοινοβούλιο να εκφέρει τη γνώμη του. Γιατί για πολλά θέματα μπορούμε να δείξουμε κοινή λογική. Και η κοινή λογική έχει μέλλον πραγματικά. Είναι ελπιδοφόρα. Και αυτό που μας λείπει μερικές φορές στα στοιχειώδη πράγματα είναι η κοινή λογική. Ο κοινό νους. Τώρα, άσχετα με τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Κορυφής, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για να είναι αυθύπαρκτο δεν θα πρέπει να γίνεται ουραγός των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων. Έχουμε μια πραγματική πολιτιστική ανέλυξη, αλλά η καθημερινότητά μας δεν δείχνει ότι στον σημερινό κόσμο θα πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλές έννοιες και σχέδια ώστε να ανταπεξέλθουμε στο ύψος των περιστάσεων και των ευθυνών μας. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Vicky. Σας ευχαριστώ. Η Βίκη απουσιάζει. Ντέρκ θα την αντικαταστήσεις, όχι. Ο Φιλίπ είναι ο επόμενος σκιώδης που είναι παρόν. Συγγνώμη που ζητώ συγγνώμη από την Αστρίντ που έλπα. Θα απαντήσω στον Ζωάν ε, Πολ στα γαλλικά, αφού μίλησε και εσύ γαλλικά θα μιλήσω και εγώ. Άκουσα ότι το ΕΡΚ σοβαρά εξετάζει την πιθανότητα της συναπόφασης και θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν μας ενδιαφέρει η μικροδιαχείριση και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Σήμερα όταν μιλούμε για ανταγωνιστικότητα, βέβαια στο πνεύμα της ε, και για το ΕΚΟΦΗΝ, ανταγωνιστικότητα σημαίνει μισθή. Εκεί περιορίζεται η ανταγωνιστικότητα για το ΕΚΟΦΗΝ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν λέω ότι η μισθή δεν είναι παράγον ε, ανταγωνιστικότητα, αλλά δεν περιορίζεται, δεν εξαντλείται η ανταγωνιστικότητα στους μισθούς. Και όταν ε, συζητάμε το Annual Growth Survey, ε, κάνουμε τη διάγνωση ότι κάποιες χώρες έχουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, αλλά η συνιστόσα της δράσης που θα πρέπει να αναλυθεί περιλαμβάνει ε, μια μισθολογική διάκριση, παρόλο που δεν είναι ακόμη κοινωτική αρμοδιότητα. Έχει μια διά, διάσταση παραγωγικότητα πόρων, ενεργειακή αποδοτικότητα κτλ. Και αν το Κοινοβούλιο καταφέρει και δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ε, τέτοιου είδους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο αξιολόγησης των ε, σχεδίων δράσης των κρατών εκεί θα είναι που θα έχουμε μια σημαντική σύμβολη, αλλά όχι μικροδιαχείριση. Λέγοντας ότι στη Γερμανία θα πρέπει να γίνει το Α, στην Πορτογαλία το Β. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά φυσικά θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι βασικές πολιτικές προϋποθέσεις προκειμένου να κάνουμε κάποιες συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αυτή θα υποβάλει στα κράτη-μέλη. Δεν μη θα υπάρχει δημοκρατική βάση για να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι πραγματικά ψηφίστηκαν αυτά τα πράγματα και εκεί θα διαπιστωθεί δημοκρατικό έλλειμμα με αποφάσεις που θα επιβάλλονται χωρίς να έχουν τη δημοκρατική νομοποίηση. Νομίζω ότι αυτό είναι το κέριο στοιχείο σήμερα και όλο και περισσότερο. Το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης είναι ζήτημα πια δημοκρατίας. Πριν μιλήσουμε για οικονομική αποτελεσματικότητα, γιατί πόρα που έχουμε από αυτή, το πρόβλημα είναι ε, θέμα δημοκρατίας. Τι νομιμότητα έχουν όλε αυτές οι διαδικασίε στα μάτια των συμπολιτών μας. Και χαίρομαι ιδιαίτερος που και το ΕΛΚ ε, είναι πρόθυμο να εξετάσει και αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι με τέτοια συζήτηση θα εκπορευθούν από το Κοινοβούλιο πιο ισορροπημένες ιδεολογικά λύσεις και πολύ πιο κοντά στο μοντέλο της ε, κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Πολύ πιο ε, ισορροπημένες από τις προτάσεις της ε, ΕΚΤ, για παράδειγμα. Φυσικά είμαστε υπέρ των προσανατολισμών της εισηγητρίας. Δεν πρόκειται να σε εγκομιάσω εδώ περισσότερο. Ελπίζω η υποστήριξη αυτή να φανεί και με έγκριση της έκθεσης στην Επιτροπή ότι αφορά τη διάκριση Ευρωζώνης και εκτός Ευρωζώνης. Σίγουρα και εκεί χρειάζονται εξελίξεις, πάντως το δικό μου μήνυμα είναι να μην ε, εμένουμε σε αυτό το διαχωρισμό. Θα δούμε ε, βέβαια το όλο το Ολυρέ στην Ευρωζώνη, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν έχουμε 17 από τη μια πλευρά και 10 από την άλλη. Έχουμε ουσιαστικά 25 και 2 ε, εκεί έγινε το διαχωρισμό σε μένα, κατά τη γνώμη μου. Γιατί με βάση τις συνθήκες δύο χώρες ε, είπαν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση ευρώ. Οι υπόλοιπε αργά ή γρήγορα θα, μάλλον θα αισθανιστούν το ευρώ. Οπότε ε, με αυτή τη λογική, με τη λογική των 25 χωρών μελών θα πρέπει να εκπονήσουμε τους μηχανισμούς οικονομικούς διακυβέρνησης. Γιατί αν κάνουμε το διαχωρισμό 17-10, είναι πραγματικά σαν να αποδεχόμαστε την αποτυχία μας και σαν να φράζουμε την περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωζώνης. Να. Οι μηχανισμοί οικονομικής διακυβέρνησης θα γίνονται με βάση τις 25 χώρες, μακάρι και τις 27. Αλλά το μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε στους 8 που έχουν, ε, που έχουν υπογράψει, να δηλαδή δεν είναι ακόμη μέσα, είναι ότι σας περιμένουμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Ευχαριστώ θεωρητικά έχουμε εξαντλήσει και αυτή τη συζήτηση ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε εκφέρει τη γνώμη μας σχετικά με το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Παρακολουθώ τον προβληματισμό της συγγήτριας και των άλλων ε, συναδέλφων που ανέδειξαν και στη σημερινή συζήτηση το θέμα της δημοκρατίας. Οι απαντήσεις που πήραμε από τη συζήτηση που έγινε πριν και με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και με τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, κατά τη γνώμη μου και νομίζω τη γνώμη και των άλλων συναδέλφων, αν κατάλαβα καλά τις τοποθετήσεις, δεν διασκέδασαν τις ανησυχίες που εκφράστηκαν ότι η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι μια άκρος αντιδημοκρατική έξω από τις συνθήκες διαδικασία και δυστυχώς η Κομισιόν και το Συμβούλιο, όπως σωστά υπογράμμισε η συγγήτρια, το αντιμετωπίζουν ως ένα διαδικαστικό θέμα και όχι ως ένα θέμα κρίσιμο, κρίσιμο πολιτικό. Η γνώμη μου επί της ουσίας είναι ότι ματαιοπονούμε να ζητάμε να καλυφθεί αυτή η έλλειψη δημοκρατίας με περισσότερο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς το Ευρωπαϊκό Εξάμενο είναι ένα στοιχείο των συνολικών πολιτικών που εκπονούνται για το ξεπέρασμα της κρίσης για την οικονομική διακυβέρνηση, που κατά τη γνώμη μου από την άποψη της πολιτικής ουσίας μας άφησε απ' έξω. Και δεν άφησα απ' έξω, δηλαδή δεν ελήφθησαν υπόψη ούτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι παρατηρήσει, ορισμένα δεν συζητήθηκαν, ούτε των Εθνικών Κοινοβουλίων και πολύ περισσότερο δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των λαών, η γνώμη των πολιτών. Θέλω να επανέλθω στι εξελίξει αυτή τη περίοδου για να σα δώσω ένα παράδειγμα. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό απελπισμένα ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα, δεν είμαι από το κυβερνητικό κόμμα, και αντιμετωπίστηκε με αυτόν τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ενώ ταυτόχρονα το αίτημα για εκλογές, εκλογές στην Ελλάδα όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, αντιμετωπίστηκε με εκβιαστικό τρόπο από την πλευρά της Κομισιόν. Ή φτιάχνετε μια κυβέρνηση, αυτά έλεγε ο κύριος Ρεν, απόψε δηλαδή για χθες, διαφορετικά δεν έχετε ούτε εκτιδώσει ούτε έβδομη, ακυρώνονται όλα είναι χαρακτηριστική και εμείς είμαστε αντιπροσωπευτικός θεσμός ότι με αφορμή και αυτά τα γεγονότα στην Ελλάδα η απέχθεια των ευρωπαϊκών θεσμών στο ζήτημα της δημοκρατίας και στο ζήτημα το να πούν οι πολίτες για μια πολιτική που τους πλήττει και η κατάσταση χειροτερεύει όλο και περισσότερο για ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα που δεν είναι μόνο πρόβλημα της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών ήδη στον ορίζοντα έχουμε την Ιταλία και τότε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα είναι χαρακτηριστική. Επομένως, συμφωνώ με τον αγώνα που γίνεται, να ακούγεται περισσότερο η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι σοβαρά θέματα, να ακούγεται η γνώμη των πολιτών, όμως όταν το απομονώνουμε αυτό καθ' αυτό, όταν το σύνολο των αποφάσεων λαμβάνονται με τέτοιο τρόπο, ε, νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε πολλά πράγματα για να είμαι, ας το πούμε έτσι, επικοδομητικός. Μια τελευταία παρατήρηση έχει σχέση με αυτό που ρώτησα τον κύριο Ρεν για όσους ήταν εδώ. Είναι φανερό ότι για να καλυφθεί αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα υπάρχουν σενάρια, τα διαβάζετε, ιδιαίτερα και από τις άλλες χώρες καταλαβαίνω με ανησυχία, περί του να τροποποιηθούν, γιατί η σημερινή συνθήκη δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία, είναι φανερό, να τροποποιηθεί η συνθήκη ούτω ώστε να προβλέπει την έξοδο ή την αποπομπή μιας χώρας από το ευρώ τέτοια σχέδια κάνουν το ευρώ εκτός των άλλων μη ελκυστικό, δεν το προστατεύουν, εισαγάγουν κενά δαιμόνια, βάζουν δηλαδή καινούρια θέματα και είναι και χαρακτηριστικοί οι χώρες, μιας και συζητάμε χώρες ευρώ μη ευρώ, οι περισσότερες χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στην Ευρωζώνη, τελευταία δείχνουν μια δυσφορία, δεν δείχνουν την επιθυμία να μπουν στη ζώνη του ευρώ. Επομένως, αυτό που μπορεί κανείς να περιμένει αν δεν αλλάξουν αυτές οι πολιτικές να έχουμε αναθεώρηση των συνθήκων που να προβλέπει πράγματα που δεν τα προβλέπει σήμερα και εκεί θα κριθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εκπρόσωπος των Ευρωπαίων πολιτών να παρέμβει πιο ουσιαστικά ούτως ώστε να αλλάξουν αυτή η λογική που ξαναλέω εκτός του ότι φορτώνει τα βάρη της κρίσης στους πολίτες είναι και έντονα αντιδημοκρατική. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Um, Η κυρία Φεραίρα επίση είναι στο κατάλογο. Αλλά προσοχή γιατί έχουμε και άλλο ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι σημαντικό. Το ζητήσαμε και τη Δευτέρα, Εκτενώ αυτό το θέμα. Παρακαλώ να είστε σύντομοι στα σχόλιά σα. Hmm. Όντως θα είμαι λακωνικότατη. Δύο σχόλια έχω μόνο. Είπα και δημοσίως ότι δεν είμαι υπέρ ούτε ενθουσιώδης ως προς την αναθεώρηση της συνθήκης αυτή τη στιγμή ειδικά. Γιατί κατά τη γνώμη μου δεν έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια ή τα όρια του ισχυρός πλαισίου εξαιτία της έλλειψης πολιτικής βούλησης. Επίσης αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμη σαφές με ποιο τρόπο αυτή, ε, θα γίνει αυτή η αλλαγή της συνθήκης, αν γίνει τελικά αυτή η αναθεώρηση. Πάντως συμφωνώ απόλυτα με τη θέση της συγκήτριας, ότι θα πρέπει να αποφανθεί το Κοινοβούλιο, ώστε το Κοινοβούλιο να καθορίσει και να οριοθετήσει τις γραμμές ε, και τα όρια της ε, δεχόμενης πιθανής αλλαγής της συνθήκης. Και είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε και διακομματική συνένεση για το θέμα αυτό. Και πραγματικά ήταν πολύ ελπιδοφόρα τα σχόλια του κυρίου Κοζές γιατί δημιουργούν προσδοκίες για την ε, πιθανή αυτή διακομματική συνένεση. Σε ό,τι αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να τον ενισχύσουμε, αλλά είναι ακόμη πιο σημαντικό το Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο να γίνει σεβαστό. Και ιδιαίτερα μια και είχαμε ευρύτατη συνένεση σε ό,τι αφορά τον ορισμό των μακροοικονομικών ανισορροπιών, ήταν ένα από τα κείμενα που έπρεπε να ψηφίσουμε στην ε, έγκριση του εξαπλού αυτού πακέτου των έξι νομοθετικών προτάσεων. Θα ήθελα να ρωτήσω αν σε επίπεδο Κοινοβουλίου ή σε επίπεδο Επιτροπής ΕΚΟΝ γίνεται μια παρακολούθηση και τι θα πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια σε σχέση με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα και αύριο στο ΕΚΟΦΗΝ. Γιατί κάποιες φήμες μας ενημερώνουν για επαναπροσδιορισμό ορισμένων θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν θέσεις που διαμορφώθηκαν μετά από πλειοψηφία και μετά από συμφωνία του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Βλέπω ότι η Πρόεδρος έφυγε και την αντικαθιστάει η Αντιπρόεδρος, αλλά εγώ θα ήθελα να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην Επιτροπή μας και να δούμε τι θα γίνει σήμερα και αύριο για το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Να μην γίνει από το Συμβούλιο μια διαφορετική ερμηνεία. Φυσικά θα ε, γίνει διάλογος και με την Επιτροπή, αλλά να μην παραγωνιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά αυτή την ερμηνεία. Για να μην παρερμηνευτούν αυτά που από κοινού είχαμε αποφασίσει και προσδιορίσει ό,τι αφορά τις ε, μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ευχαριστώ. Um, okay, thank you. Ευχαριστώ. Κύριε Μπερές, να σας ξαναδώσω το λόγο εν συντομία για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση γιατί έχουμε χρονικό περιορισμό. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφου του οποίους άκουσα με μεγάλη προσοχή. Δύο λόγια όσον αφορά το θέμα της συναπόφαση. Γιατί θα είναι και η πιο σημαντική απόφαση που θα πάρουμε εφόσον ακολουθήσουμε βέβαια τις προτάσει που κάνω. Βεβαιώ δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πεπατημένη σε μια τέτοια περίπτωση, σαν αυτή δηλαδή που παρουσιάζεται σήμερα μπροστά μας. Αλλά ε, έχουμε εφαρμόσει μια σχετική διαδικασία συναπόφασης ε, την προηγούμενη φορά για τις προοπτικές. Ε, δεν κράτησε τρεις μήνες, ήταν λίγο παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι με λίγη καλή θέληση έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Και εξάλλου, έτσι πιέζοντας ε, θα βελτιώσουμε τα πράγματα, γιατί και εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να πιέσουμε τους εαυτούς μας έτσι ώστε να βελτιωθούμε, να αλλάξουμε τις συνήθειές μας κτλ. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι θα πρέπει να έχουμε και υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Να σας θυμίσω ότι θα ψηφίσουμε τη Δευτέρα του Στρασβούργου για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους ε, συνέβαλαν. Ε, θα πρέπει τώρα να στραφώ προς τον συνάδελφο Σικλούνα. Τελευταίο σημείο, γιατί και εγώ θα πρέπει να φύγω. Το ενωσιακό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης ο κύριος Φόξ, ο εισηγητής δεν είναι εδώ, αλλά φαίνεται ότι θα πάρει τον, το λόγο στη θέση του. Ναι. Το τρένο του κυρίου Φόξ καθυστέρησε. Θα διαβάσω τις σημειώσεις του. Πρώτα απ' όλα καλωσορίζει την πράσινη βίβλο της Κομισιόν για ένα πλαίσιο εταιρική διακυβέρνησης ε, με τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Μετά την οικονομική κρίση ήταν σαφές πως ε, κάποιες ρυθμιστικές αλλαγές ήταν απαραίτητες στις αγορές μας και στις εταιρείε μας. Όμως η αλλαγή αυτή πρέπει να είναι αναλογική. Όταν εξετάζουμε το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να διαχωρίσουμε από την προσέγγιση μεγάλων συστημικά σημαντικών εταιριών και των υπολείπων ανωνύμων εταιριών. Όταν υιοθετήσαμε τη σχετική έκθεση για, τα, για τους χρηματοοικονομικούς οίκους. Η Κομισιόν σωστά είπε πως θα πρέπει βάση της προσέγγισής μας να είναι η αναλογικότητα. Η ποικιλία των διαφόρων δομών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ποικιλία των προσεγγίσεων των ε, κρατών μελών στην ρύθμιση και το να αναγνωρίσουμε πως μία ενιαία προσέγγιση δεν ε, θα ωφελήσει την ανταγωνιστικότητα των ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι σημαντική εάν συμφωνούμε πως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να τηρούν υψηλότερες προδιαγραφές λόγω της συστημικής τους φύσης. Τότε προκύπτει πως οι υπόλοιπες εταιρείες θα πρέπει να έχουν ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον. Δεν θα πρέπει να βλάψουμε την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιριών με ε, ρυθμίσει οι οποίε δεν χρειάζονται. Η βασική επιτροπή είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εμεί έχουμε περιορισμένη αρμοδιότητα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στου συγκεκριμένου αυτού τομεί. Η ε, γενική προσέγγιση του κυρίου Φόξ είναι η εξή σεβασμό για το υπάρχον πλαίσιο για τις διάφορες εισηγμένες εταιρείες. Επίσης να προσπαθήσουμε να βρίσουμε ένα πλαίσιο έτσι ώστε να είναι υπόλογε στου μετόχου οι εταιρείε, να δούμε τι βέλτιστε πρακτικέ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να απτυχθεί ένα κώδικα συμπεριφορά που να το αντικατοπτρίζει. Ο ρόλο των μετόχων θα πρέπει να ενισχυθεί, ειδικά όσον αφορά τον έλεγχο των εταιριών. Θα πρέπει να ενημερώνουν επίση τι ρυθμιστικέ αρχέ όταν αποκλίνει από τον κώδικα χωρί ιδιαίτερο λόγο μια εταιρεία. Επίσης το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τους θεσμικούς επενδυτές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια νομοθεσία για να αποφευχθεί η λογική των βραχυχρόνιων κερδών. Επίσης θα συνεργαστούμε με τον κύριο Μπόντου για να ληφθεί υπόψη η άποψη της Επιτροπής μας και αναμένει και τις απόψεις των υπολείπων συναδέλφων, ιδιαίτερα των σχεδόν. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ. Τώρα κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή μα τον κύριο Φόξ, για την γνωμοδότησή του και χαίρομαι που εξετάζουμε αυτό το θέμα, μια και είναι πολύ χρήσιμη η συζήτηση αυτή για την εταιρική διακυβέρνηση. Γιατί έτσι θα βελτιώσουμε και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Συμφωνώ με τον εισηγητή μας ότι το θέμα είναι λεπτό και ευαίσθητο. Γιατί μερικοί από τους κανονισμούς ε, ε, εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα, δεν είναι κοινωτική αρμοδιότητα και άρα δεν μπορούμε να έχουμε κοινούς κοινωτικούς κανόνες. Πάντως, ε, όταν εξετάζουμε ένα θέμα, η κοινή γνώμη είναι στραμμένη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιμένει λύση. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία θέματα. Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχη και οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. Καταρχήν, το Διοικητικό Συμβούλιο. Ε, το θέμα αυτό το αναφέρει ο ο εισηγητής. Είναι σημαντικό βέβαια το θέμα της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Πολύ πιο σημαντικό είναι όμως να αποφύγουμε τη σώρευση της γραφειοκρατίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν μπορούμε να διαφοροποιήσουμε κάπως τη θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά το θέμα των εταιριών που δεν είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο και που παρόλα αυτά έχουν τεράστιο οικονομικό δυναμικό, αλλά δεν υπάγονται σε ρυθμίσεις ε, ε, ως προς τη λειτουργία τους. Ο κύριος Φόξ προσέγγισε αυτό το θέμα από το πρίσμα του κώδικα, αλλά η προσέγγιση αυτή θα είναι σωστή μόνο εφόσον δεν ε, έρθει σε αντίθεση με άλλους κανόνες της εσωτερικής αγοράς ή καταστρατηγήσει συμφέροντα άλλων φορέων. Ένα άλλο ζήτημα προς εξέταση είναι το κατά πόσο η εταιρική διακυβέρνηση η εταιρική διαχείριση θα μπορούσε να συνοδευτεί από εποπτεία κρατική ή από εξωτερική αξιολόγηση. Νομίζω ότι καλό θα είναι να αποφύγουμε αυτό το θέμα. Η πράσινη βίβλος αναφέρει και το θέμα της ε, ισότητας των δύο φύλων ό,τι αφορά την εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το θέμα αυτό δεν νομίζω ότι είναι το σημαντικό, γιατί δεν είναι σημαντικό το θέμα της ισότητας των φύλων, αλλά γιατί αποσπά την προσοχή μας από πιο σημαντικά ζητήματα. Ανακεφαλαιώνοντας, ήθελα να πω ότι μία αποτελεσματική εταιρική διαχείριση και ένα σύστημα που θα την εξασφαλίζει είναι ε, χρήσιμα και τα κριτήρια αυτής της ε, εταιρική διακυβέρνησης θα πρέπει να προσδιορίζονται εκ των προτέρων και να είναι υπόλογο το Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης είναι σημαντικό ότι αυτά τα μέτρα που είναι σημαντικό τα μέτρα που θα προτείνει η έκθεση να λαμβάνουν υπόψη και την ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας και όχι ενίσχυσης της. Η πράσινη βίβλος ε, θέτει κάποιους στόχους, αλλά αποφεύγει την αναφορά των μέτρων με τα οποία θα υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί. Εμείς στις τροπολογίες μας ε, θα αναφερθούμε σε όλα αυτά τα θέματα και θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ τον συντάκτη της γνωμοδότησης για το πόνημά του. Σας ευχαριστώ, είμαι ο ε, των Σοσιαλδημοκρατών και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φόξ για τις ενδιαφέρουσες ε, προτάσεις του που αποτελούν βάση καλή έκθεσης. Πράγματι, θα πρέπει να δούμε με ευέλικτο τρόπο την εταιρική διακυβέρνηση με ιδιαίτερο βάρος μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλωσορίζω τις παρατηρήσεις του εισηγητή που ενσωματώνουν τις προτάσεις της Κομισιόν για κατάργηση των υποχρεώσεων αναφοράς κάθε τρίμηνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμφωνώ επίσης μαζί του για τον κώδικα συμπεριφοράς. what the success of Όσον αφορά αυτό το οποίο ονομάζει επιτυχία του Comply and Explain, μπορεί να είναι ένας λογικό κανόνα αρκεί να δίνουν λεπτομερείς εξηγήσει οι εταιρείε ακόμα και όταν σκοπεύουν να αποκλίνουν από τον κώδικα. Η πράσινη βίβλος της Κομισιόν εξετάζει ευρήματα μελετών παρακολούθησης της ε, εταιρική διακυβέρνησης και διαπιστώνει διάφορες ελλείψεις. Και βεβαίως εδώ να επιστήσω την προσοχή σας στον Σουηδικό κώδικα που απαιτεί από τις κυβερνήσεις, από τις επιχειρήσεις να πούν σε ποιου κανόνε δεν συμμορφώθηκαν και τι σκοπεύουν να κάνουν γι' αυτό. Αυτό είναι καλύτερο. Επίση, χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι βλέπω στην πράσινη βίβλο το ότι θα πρέπει οι εταιρείε ε, να αναφέρουν την πολιτική τους και την αμοιβή των ε, διευθυντών τους και το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών για την αμοιβή των διευθυντών τους. Έτσι αυξηθεί η διαφάνεια και θα μειωθεί η αναντιστοιχεία μεταξύ πληρωμών στελεχών και απόδοσης εταιρεία. Επίσης, ε, το σημαντικό ρόλο των μετόχων, ε, τα δικαιώματα ψήφου και συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν να αυξηθεί η ταυτοποίηση των μετόχων. Τέλος, να προτείνω κάποιες τροπολογίες για την ιδιοκτησία από του εργαζόμενου που βλέπουν πως αυξάνεται την παραγωγικότητα και μειώνει τι κοινωνικές εντάσει. Θα ήθελα επίσης να επεκτείνουν και να ενθαρρύνουν τέτοια ιδιοκτησία τα κράτη-μέλη μέσω εθνικών φορολογικών βασότων. From the Greek, Ο Σβέν από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. just replacing our shadow. Αντικαθιστώ το μας. Να σας κάνω κάποια σχόλια. Ε, όλοι κάποιον αντικαθιστούμε εδώ πέρα, μόνο ο πρόεδρος έχει μείνει. Κάποια πραγματάκια. Πρώτα, προφανώς, υπάρχουν κάποιες εντάσεις. Πρώτα, έχουμε μία αρχή εμείς, μία προτίμηση μάλλον, εκεί όπου δεν λειτουργεί αποτελεσματικά η προαιρετική νομοθεσία να περάσουμε σε ε, νομοθεσία κανονική. Σαφώς η γνωμοδότηση Κάρας είναι σημαντική, τη στηρίζουμε εκεί που λέει πως αναγνωρίζει πως η οικονομική κρίση θα οδηγήσει σε έλλειψη αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων αρχών ε, εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεραίνει πως ε, απαιτούνται κάποιες ε, νομικά δεσμευτικές ρήτρες και κάποια προαιρετική, κάποιες προαιρετικές ρυθμίσεις. Όσον αφορά τώρα την αμοιβή των στελεχών, ιδιαίτερα στα υψηλότερα κλιμάκια, ζητά περισσότερη διαφάνεια και δεσμευτικούς κανόνες για να καλυφθεί η ψαλίδα μεταξύ αμοιβή και δημιουργίας αξίας ιδιαίτερα, αλλά χωρίς να περιορίζεται, στο χρηματοοικονομικό τομέα. στη συζήτηση για, το, για τα φύλλα θεωρούμε πως η αποτελεσματική προσέγγιση της Νορβηγίας θα πρέπει να στηριχτεί και να υπάρξει μια ισορροπία των φίλων στα διοικητικά συμβούλια καθώς βλέπουμε πως αυτό δεν γίνεται μόνο με τα προαιρετικά μέτρα και Πέρα από αυτό θεωρούμε πως υπάρχει εδώ πέρα βεβαίως μια προτίμηση προς τους ε, μετόχους και ε, βεβαίως η εταιρική διακυβέρνηση δεν ε, είναι μόνο το συμφέρον των μετόχων. Θεωρούμε πως πρέπει να έχουν περισσότερη δύναμη οι μέτοχοι στις εταιρείες και να συνεισφέρουν σε πιο υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση. Και βεβαίω εδώ πέρα δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για μετόχους, αλλά για όλους τους ενδιαφερόμενους. ΜΚΟ, περιβαλλοντικές οργανώσεις θα πρέπει να είναι σε μια θέση να αξιολογήσουν το εάν η διακυβέρνηση αυτή συμφωνεί με το μακροπρόθεσμο της εταιρείας, κάτι το οποίο σημαίνει περισσότερη διαφάνεια, ειδικά για τις μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή να συμπεριληφθούν ενδιαφερόμενοι είναι και στο μακροπρόθεσμο, ε, προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων. Και θεωρούμε πως ε, με βάση αυτά τα οποία έχει πει ο εισηγητής πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις για να γίνει η γνωμοδότηση ε, πιο ισορροπημένη. Ευχαριστώ. Σας έχει απομείνει μόνο ένα δίλεπτο. Ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι θα διαβιβάσω τις παρατηρήσεις και τις δικές σας και των συναδέλφων στον συντάκτη της γνωμοδότης. Ιδιαίτερα οι παρατηρήσεις του κυρίου Google, Google δίνουν τροφή για σκέψη και σίγουρα ε, στόχος του συγκεκριτού δεν είναι η μικροδιαχείριση των επιχειρήσεων εκ των άνω. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζητούμενο της γνωμοδότησης αλλά για περισσότερε λεπτομέρειε παραπέμπω σε προσωπική επαφή με τον εισηγητή τον κύριο Φόξ. Ωραία. Το χρονοδιάγραμμα μα τώρα για την γνωμοδότηση. Προθεσμία για τι τροπολογίε ε, λίγη στι 15 Νοεμβρίου το μεσημέρι. Εξέταση τροπολογιών στις 29 Νοεμβρίου. Ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ 19 Δεκεμβρίου και ψηφοφορία στην Αρμόδια Κατουσία Επιτροπή που είναι η Γιούρε, η νομική είναι στις 26 Ιανουαρίου για να περάσει η έκθεση στην Ολομέλεια του Μαρτίου, στην, στην πρώτη. Η επόμενη μας συνεδρίαση, Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Λίγη συνεδρίαση.